Chers collègues, je vous propose de euh, recommencer. Ας ξεκινήσουμε, τη οι συνάδελφοι, αν θέλει αυτό, τις εργασίες μας. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, γιατί θα πρέπει, εφόσον βρισκόμαστε στην αρχή της ε, δεύτερης, ε, του δεύτερου μισού της θητείας μας και στην αρχή του 2012, πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, να ξεκινήσουμε μέσα στο πρόγραμμα εργασιών μας με τους αποκεκεντρωμένους φορείς Είμαστε μια επιτροπή με πολλά πλούτη. Γιατί έχουμε αποκεντρωμένους φορείς, ένα κέντρο και ένα καταπίστευμα που εξαρτώνται από την επιτροπή μας. Η εμπειρογνωμοσύνη λοιπόν την οποία έχουμε αποκτήσει και αποκτούμε κάθε μέρα θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τα θέματα της αρμοδιότητας και του ενδιαφέροντος της Επιτροπής μας και τα οποία συνδέονται με πολλά διακυβευόμενα. Βάση της παγίας πρακτικής που οι παλιότεροι γνωρίζουν, θα δώσω σε όλους σας τη δυνατότητα να κάνετε μια παρέμβαση η οποία θα είναι ίσως κάπως ματαιωτικού χαρακτήρα γιατί αναφέρεστε στην Επιτροπή μας, αλλά μόνο για 6 με 8 λεπτά ο καθένας, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ως το δυνατόν πλέον καρποφορότερη. Με τον πιο γραφειοκρατικό τρόπο λοιπόν θα δώσω το λόγο στη σειρά την αλφαβητική στους εκπροσώπους των φορέων, βάσει αλφαβητική σειρά των φορέων Δίνω το λόγο στην κυρία Χρήστα Σέτλατσεκ για τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να ακούσουμε πρώτα όλες τις παρεμβάσεις και μετά στο τέλος να γίνουν οι παρατηρήσεις. Γιατί αν σταματάμε κάθε φορά σε κάθε φορέα, τότε θα ξεχάσουμε. Θα χάσουμε το οδηγό νήμα. Κύριε Σέντλατσεκ, έχετε το λόγο να παρουσιάσετε το φορέα σα. 6-7 λεπτά. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθουμε να σας πληροφορήσουμε για την περσινή μας εργασία και για τα σχέδιά μας για εφέτος. Έχετε στους φακέλους σας μπροστά σας ελπίζω τα κύρια στοιχεία του προγράμματός μας καθώς και την πιο λεπτομερή επεξεργασία του για το 12. Γι' αυτό ακροθυγός μόνο θα αναφέρω τα κυριότερα και αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις με χαρά να τις απαντήσω. Ε? Συνεχίζουμε να χορηγούμε πληροφόρηση και στήριξη σε εταιρείε και εργαζόμενους ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν για να παραμείνουν οι τόποι εργασίας ασφαλείς και υγιείς. Επίσης συνεννοούμαστε με λήπτες αποφάσεων στους δύσκολους καιρούς της μεγάλης ανεργίας που παρατηρούμε και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν τον πειρασμό να βάλουν την οικονομική αποτελεσματικότητα πάνω από την ίδια τους την υγεία και την ευημερία για να κρατήσουν τη δουλειά τους πάση θυσία ακόμη και εναντίον της υγείας των. Τα μέτρα λιτότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη το τονίζουν αυτό ακόμη περισσότερο το χειροτερεύουν. Είναι πολύ μειοπική αυτή η προσέγγιση και σε λίγο θα δούμε τα ικτρά αποτελέσματα του λάθους αυτού και, και στην οικονομία και στην επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών και στην υγεία. Για όποιον δεν πείθεται να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα. Δείγματα. Το 10 δημοσιεύσαμε μια ευρωπαϊκή μελέτη επιχειρήσεων καινούριων επιχειρήσεων που ήταν η πρώτη του είδους της για την υγεία στους τόπους εργασίας. Μάθαμε πολλά από αυτή τη μελέτη. Εξετάζοντας γενικά την κατάσταση της υγείας στους τόπους εργασίας. Μάθαμε τους λόγους για τους οποίους η αξιολόγηση των κινδύνων πολλές φορές δεν είχαν γίνει ποτέ. Ουδέποτε. Δηλαδή ανακαλύψαμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται τη βοήθειά μας και συνεχίζουμε να κάνουμε προσπάθειες για να τη χορηγήσουμε αυτή τη βοήθεια. Το 12 θα γράψουμε πιο λεπτομερείς μελέτες με βάση τις αναλύσεις μας. Μέχρι τώρα, όχι μόνο στην έδρα μας στον Μπιλμπάο αλλά και αλλού, οι πληροφορίες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί γενικώ από διάφορους ηγέτες επιχειρήσεων και πολιτικούς. Πώς χρησιμοποιούνται στην πράξη τα συμπαράσματά μας. Η αξιολόγησή μας γίνεται συνεχώς και online και την λέμε όιρα. Και ε, είναι άμεσο αποτέλεσμα των συμπερασμάτων της μελέτης μας για τις μικρόμεσες και πολύ μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σε ευρωπαϊκούς κύκλους ακούγεται πολλή συζήτηση που αμφισβητεί την ανάγκη αξιολόγησης κινδύνων στον τόπο εργασίας και που θέτει το ερώτημα μήπως δεν είναι καμιά άχρηστη επιβάρυνση των επιχειρήσεων αυτή η αξιολόγηση. Τώρα όμως γνωρίζουμε ότι μια σωστή αξιολόγηση του κινδύνου είναι ο κρογωνιαίος λίθος της σωστής υγειονομικής διαχείρισης. Γι' αυτό αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο που είναι εύχριστο δεν βοηθάει μόνο τις επιχειρήσεις να πληρούν τους όρους που τους έχουν τεθεί, αλλά επίσης αυτόματα γράφει και εκθέσεις μόλις λάβει τα, τα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε είμαστε σίγουροι ότι οι αξιολογήσεις γίνονται όπως πρέπει με γραπτά στοιχεία που βασίζονται σε ένα πρότυπο που πρωτοεφάρμοσε η Ολλανδική κυβέρνηση. Και έχουμε 100, ε, στην Ολλανδία έχουν 150 συγκεκριμένες εφαρμογές του ανατομέα. Επίσης, δείχνει στο σελίδα μας πόσο συμμετέχει και ο ίδιος ο εργαζόμενος σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η επόμενη διετής καμπάνια μας θα αναφέρεται σε δύο κύρια θέματα, τη συμμετοχή των εργαζομένων και την βελτίωση των ελέγχων. Αυτά είναι τα δύο μαγικά συστατικά. Η καμπάνια αυτή θα αρχίσει τον Απρίλιο και αναγνωρίζεται ήδη ως η μεγαλύτερη παγκόσμια καμπάνια του είδους της. Συμπεριλαμβάνει περισσότερες χώρες από ποτέ και θα διαρκέσει όπως είπα δύο χρόνια, γι' αυτό είναι διετής. Great and the Κάνουμε και προβλέψεις για την εμφάνιση πιθανών νέων κινδύνων με την χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας. Και σας το λέω ειλικρινά, κανείς δεν μας έχει επικρίνει για την προώθησή μας του λεγόμενου πρασίνου τομέα. Αλλά πρέπει να δοθεί ιδέουσα προσοχή, ιδέουσα προσοχή να μειωθεί και αν γίνεται και να καταργηθούν τέτοιοι κίνδυνοι. Ό,τι είναι πράσινο δεν είναι κατά ανάγκη και ασφαλές. Αλλά η σωστή γνώση του κινδύνου είναι. Και η δική μας προσέγγιση είναι να δίνουμε ολόκληρη εργαλειοθήκη στις επιχειρήσεις με τις πληροφορίες που τους διαθέτουμε και μάλιστα με πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων, πληροφοριακών προϊόντων. Εκτός από τα παραδείγματα αυτά υποστηρίζουμε και το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γυράνσεως. Για να, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να παραμείνουν υγιείς μέχρι την ημέρα της συνταξιοδοτήσεώς του και παραπέρα. η πρόορη απόσυρση των εργαζομένων από τον τόπο εργασίας λόγω όλο και περισσότερων αναπηριών είναι κάτι που πλήττει σοβαρά το περιβάλλον εργασίας γιατί υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι η υγιής παραμονή των εργαζομένων στους τόπους εργασίας είναι βιώσιμος τρόπος ανάπτυξης. Και αν χρειαστεί, αν συμβεί να αρρωστήσουν ή να ατυχήσουν, να πάθουν ατυχήματα δηλαδή, πρέπει να είναι σε θέση μετά να επιστρέφουν υγιείς στην εργασία τους, υγιέστεροι από πριν. Τέλος, πρέπει να παραμείνουμε να διατηρήσουμε ένα κριτικό πνεύμα ως προς τα επιτεύγματά μας και την θέση μας στο σημερινό πολιτικό και οικονομικό κλίμα. Η συμβολή μας στην επίτευξη των στόχων του 20 είναι η καταλληλότερη γι' αυτό μέθοδος. Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο ανέλαβα τα καθήκοντά μου, θέλησαν να αρχίσει μια στρατηγική, ένα στρατηγικό σχεδιασμός μέσα στα πλαίσια του Διοικητικού μας Συμβουλίου που αποτελείται από κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενους καθώς και με το υπόλοιπο πυροσωπικό. Αυτό συνεχίζεται και φέτος και με μεγάλη χαρά ελπίζω να είμαι σε θέση να σας πω καλά νέα μόλις το καταφέρουμε θέλουμε να παραμείνουμε We need to listen to our... κέντρο αρι, αριστείας. Γιατί στα ταραγμένα αυτά νερά πρέπει να μπορούν οι εργαζόμενοι κάπου να κουμπίσουν. Πρέπει να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν εφόσον το αγνοούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας επίτευγμα, δηλαδή προσφέρουμε πολλά. Προσβλέπω στην τακτική συνεννόηση μαζί σας, γιατί ελπίζω να με καλείτε συχνά στην Επιτροπή Απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, διότι η συνεχιζόμενη υποστήριξή σας έχουν ήδη υπάρξει μία έμπνευση για μας, για την οποία σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας που ήταν εμπεριστατωμένη σε σχέση με, τα, με τις προσπάθειες που καταβάλλετε για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Περνάμε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. Δίνω το λόγο στον κύριο Κριστιαν Λετμάιερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Μπερές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμα ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο μας στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ενημέρωση που σας έχουμε δώσει και σε άλλα πληροφοριακά έγγραφα τα οποία απεστάλησαν σε εσά πρόσφατα σε σχέση με τις προσπάθειες για να διαμορφωθεί καλύτερα η διαβίου ανάπτυξης για μια πληρέστερη παρουσίαση του ΣΕΔΕΦΟΠ του παρελθόντος του και του μέλλοντος. Σας παραπέμπω στην ετήσια έκθεση του 2011 που θα είναι διαθέσιμη σύντομα και επίσης τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές μας που επίσης θα διατυπωθούν εν καιρό. Πάνω από 150 συνδιασκέψεων οργάνωσε, συνδιοργάνωσε το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. 108 συναντήσεις ή εργαστήρια και το έργο μας όλο και περισσότερο αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο σε έγγραφα εργασίας και πολιτικής πέραν αυτών των παραπομπών σε επιστημονικά περιοδικά που καταδεικνύει ότι ο αντίκτυπος της δουλειάς μας αυξάνεται και ότι ο στόχος μας να γίνουμε μια έγκυρη πηγή για τα θέματα των προσόντων και της διαβίου μάθησης είναι στο δρόμο της επίτευξης. Είναι μια επιτυχία η οποία χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπαθίες μας. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει εφαρμόσει πλήρως τον προϋπολογισμό του 2011 που καταδεικνύει την καλύτερη σχεδίαση, την καλύτερη παρακολούθηση, χάρη και στα δικά σας σχόλια. Έχουμε μελλοντικό χώρο και για περαιτέρω βελτίωση. Πιστεύω πρέπει να βελτιώσουμε καλύτερα τη σχέση μας με τα μέσα ενημέρωσης, να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση για την ανάγκη της διαβίου μάθησης και την ανάγκη να τονιστεί αυτό στις τωρινές εξελίξεις. Το 12 το ΣΕΔΕΦΟΠ θα συνεχίσει να αναπτύσσει εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει προχωρήσει σημαντικά η εκπόνηση αυτών των εργαλείων σε ό,τι αφορά το εθνικό πλαίσιο πιστοποίησης με την ε, εφαρμογή του συστήματος EasyNet για την επαγγελματική ε, εκπαίδευση και επιστοποίησή της που βρίσκεται σε ένα εμβριακό ακόμα στάδιο. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν για την επιστοποίηση και η ποιοτική εξασφάλιση, η εγγύηση ασφάλειας είναι σημαντικά εργαλεία. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνέργεια σε εθνικό επίπεδο και συμβατότητα, αλλά συγχρόνως και συνεκτικότητα και συνεκρισιμότητα μεταξύ κρατών μερών. Το Europass ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τα βιογραφικά τα οποία είναι επιγραμμικού χαρακτήρα. Αλλά για να γίνουν πιο ορατά τα άτυπα, τα αποτελέσματα άτυπης μάθησης χρειάζονται και περαιτέρω βελτιώσεις. Αυτό θα βοηθήσει και την καλύτερη λειτουργία του EasyWeb και του μηχανισμού επαλήθευσης. Αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω όμως είναι η ανάγκη να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα εργαλεία με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι κομβικό αυτό αν θέλουμε να κάνουμε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο εύκαμπτα και να δώσουμε τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να μετακινούνται από διάφορες μορφές κατάρτισης και παιδείας και φυσικά και χώρων εργασίας. Δεν είναι κάτι τετριμένο, δεν είναι κάτι εύκολο. Το σούτορ μάλλον καθώς χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και συνεκρισιμότητα μεταξύ εθνικών συστημάτων. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ παρακολουθεί τη λεγόμενη διαδικασία αναφοράς και υποστηρίζει τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό, γιατί αυτά τα βήματα θα βοηθήσουν την διαπερατότητα και την ευελιξία των συστημάτων κατάρτισης και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να έχουμε και περισσότερη εστίαση στην εμπειρία που κάτω κατά την εργασία και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη αναβάθμιση των προσόντων μιας γυράσκουσας εργατικής δύναμης για να υπάρχει καλύτερη προσαρμογή των προσόντων τους προς τις ανάγκες της αγοράς. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες ανισομέρειες στην αγορά εργασίας Ιδίω την μεγάλη ανεργία των νέων και τη μεγάλη ανεργία γέννη, ιδίω σε χώρες οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την χρηματοοικονομική κρίση. Αυτό έδειξε ότι υπήρξαν κάποιες πρακτικές οι οποίες ήταν μη βιώσιμες σε μακροοικονομικό επίπεδο και οδήγησε σε ύφεση. Ακόμα και αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πάντα να βρίσκουν άτομα με τα κατάλληλα προσόντα και πολλοί απόφοιτοι με υψηλά προσόντα παίρνουν θέσει εργασία που είναι κάτω από το επίπεδό του. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει σωστή συνάρμοση των προσόντων με τι ανάγκε είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και την ποιότητα της εργασίας αλλά και την προσωπική αντίληψη της ποιότητας της εργασίας και την ευμάρεια. Το ΣΕΔΕΦΟΠ εργάζεται για να εντοπίσει τις ανάγκες δεξιοτήτων και να βρει πόσο μεγάλη είναι η ανισομέρεια μεταξύ προσόντων και θέσεων εργασίας που δεν είναι μονάχα οξία αυτή η ανισομέρεια σε εποχές κρίσης, αλλά εξακολουθεί να περιμένει και σε καλύτερες εποχές. Θα πρέπει η έρευνα αυτή για τα προσόντα να οδηγήσει σε μια καλύτερη και τελευρύτερη συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ό,τι ξέρουμε λοιπόν για τις για τα προσόντα θα πρέπει να μεταφραστεί σε τροποποίηση στα συστήματα εκπαίδευσης για να προσαρμόσουμε την παροχή, την προσφορά με την ζήτηση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να, να κατευθύνουμε καλύτερα τους νέους σε επιλογή καριέρας ή εκπαίδευσης ή και κατάρτισης. Όλα αυτά σημαίνουν να υπάρξει μια ολοκλήρωση των στοιχείων πληροφορίας και να εξαλείψουμε τις τις ανισομέρειες σε ό,τι αφορά τις ε, αποκτήσεις προσόντων για την διαβίου ε, εκπαίδευση. Επίσης πρέπει να είναι ανοιχτά και ευέλικτα τα συστήματα για να μπορούν τα άτομα να προσαρμόσουν καλύτερα τις ε, δεξιότητές τους στις ανάγκες τους. Όλα αυτά νομίζω ότι καταδεικνύουν ότι το Σέντεφοπ αντιμετωπίζει θέματα άμεσης σημασίας για την ευρωπαϊκή πολιτική και εμπλέκονται και οι εθνικές κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι σε όλο αυτό το προβληματισμό. Οι μεσοπρόθεσμες μας προτεραιότητες έχουν σαν στόχο να εστιάσουμε καλύτερα στις πιο έντονες προκλήσεις μέσα στο τωρινό ζωφερό οικονομικό κλίμα. Ελπίζω ότι μπόρεσα να σας δείξω ότι το έργο μας αφορά αλληλένδετους και διασυνδεδεμένους κλάδους και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ τους που είναι ουσιώδεις για να μπορέσει ο κάθε κλάδος να αναπτύξει την πλήρη δυναμικότητά του χάρη στην καταπληκτική εργασία των εμπειρογνώμονων του ΣΕΔΕΦΟΠ, ζητήσαμε να πάρουμε και περαιτέρω καθήκοντα. Είτε, παραδείγματος χάρη, την ε, διαδικασία της Κοπελχάγης για τις πρακτικές εργασίες, όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν Plus, ή επίσης το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων που θα επιτρέψει την καταγραφή και τεκμηρίωση μη τυπικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί ή επίσης να παρακολουθήσει την εξέλιξη των προσόντων και να βοηθήσει την ανάπτυξη του ΕΣΚΟ που συσχετίζει τα προσόντα όπως αναφέρονται στα προγράμματα μαθημάτων με προσόντα για διάφορα επαγγέλματα όπως τα ορίζει η αγορά εργασίας. Εν τέλει θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τα έργα ανακαίνησης και αποκατασκευής του κτιρίου του ΣΕΔΕΦΟΠ βάσει προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2011 και αν πάνε όλα καλά θα έχουν περατωθεί εργασίες τον Ιούνιο του 2011 θα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και πάλι τις ε, εγκαταστάσεις διασκέψεων στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, όπως ξέρουν περισσότεροι από εσά, η πρώτη διαδικασία πρόσληψης για ένα νέο διευθυντή του ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2011 και θα καταλήξει, ελπίζουμε, τον Ιούνιο του 2012. Επομένως θα έχει ένα νέο διευθυντή το κέντρο, κατά πάσα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, αν θέλει ο Θεός. Όπως όλοι οι αποκεντρωμένοι φορείς, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ θα θέλει από το 2013 να αντιμετωπίσει μια υποχρεωτική μείωση προσωπικού και ένα προϋπολογισμό μηδενικής αύξησης. Τα τελευταία χρόνια το κέντρο μας έχει ακολουθήσει μια πολιτική αυξανόμενη αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και έχει εστιάσει την προσοχή του σε θέματα μεγάλης προτεραιότητας, νομίζω ότι αυτή η πρόσθετη απέτηση θα περιορίσει σημαντικά σχέδια τα οποία μπορεί να χρειαστεί να αναβληθούν ή να ακυρωθούν παραγωγικά η συνεισφορά μας σε συνδιασκέψεις και συζητήσεις δημοσίου χαρακτήρα θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο <clears throat> και ιδίω την Επιτροπή Απασχόλησης για την υποστήριξή σας και για την καλή συνεργασία που έχετε, είχατε μαζί μας στο παρελθόν και σας ζητώ να συνεχίσετε αυτή την υποστήριξη και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών διαβίωση και εργασία. Ο κύριος Μενέντες Βάλτες έχει το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι το δεύτερο μου έτος εδώ. Πέρσι μόλις ένα μήνα είχα που είχα αναλάβει τα καθήκοντά μου όταν παρουσιάστηκα εδώ. Τώρα περισσότερο πείρα πρέπει να έχω. Να σα παρουσιάσω κάποια επιτεύγματα του προγράμματο εργασία ε, του 2011 και κάποια στοιχεία του προγράμματο 2012. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε γιατί έχετε λάβει ε, σύνοψη των προγραμμάτων εργασία. Αυτά τα δύο χρόνια, 2011 και 2012, θα είναι τα δύο τελικά χρόνια του ισχύοντος τετραετού προγράμματο που έχει τίτλο «Η Ευρώπη στη δουλειά, ε, δυνατότητε για όλου, Προσπαθούμε να εκπληρώσουμε ε, το ρόλο τη υπηρεσία μα που έχει τριπλό στόχο να διαδώσει τη γνώση σε εκεί στο υπουργό τη πολιτική στον τομέα κοινωνική πολιτική και απασχόληση με περιορισμένο προπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ χωρί να αυξήσουμε ανθρωπίνους πόρου και θέλουμε να προσαρμοστούμε στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν συντάσαμε το παρόν τετραετές ε, πρόγραμμα ε, δεν είχε ξεκινήσει η κρίση. Το 2011 καλύψαμε πάνω από το 99% του προπολογισμού, δημοσιεύσαμε πάνω από 180 δημοσιεύματα και στις διάφορες γλώσσες πάνω από χίλιες εκθέσεις. Ε, εκτυπώθηκαν ή παρουσιάστηκαν στη σελίδα μας και κάποιοι δείκτες επιδόσεων μας δείχνουν πώς χρησιμοποιούν ενδιαφερόμενοι η τεχνογνωσία μας. Πάνω από 118.000 ε, ε, εκθέσεις κατέβηκαν στη σελίδα μας ε, που αφορούσαν ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολίτες πάνω από 330.000 ε, επαφές για την αριστεία πάνω από 450 παραθέσεις σε επιστημονικά έγγραφα και εκδόσεις. Και αυτό και πάνω από 170 παραθέσει από εκείνου που διαμορφώνουν πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για διαμόρφωση πολιτική. Ξεκινήσαμε τώρα τι συζητήσει του επόμενου τετραετούς προγράμματο, 2013 με 2016. Γίνονται σε πολλαπλά επίπεδα διαβουλεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι η Δημοσιονομική Αρχή θα συμμετάσχει και οι κυβερνήσει θα συμμετάσχουν και εργοδότες και εργαζόμενοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Και θα παρουσιάσουμε το αργότερο Ιανουάριο του 2013 το νέο μας πρόγραμμα, τετραετές πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι έρευνες μας α, βασιζόταν σε πολιτική κυρίως. Βασικές δραστηριότητες ήταν και θα είναι οι ευρωπαϊκοί, ε, ευρωπαϊκές έρευνες που διεξάγουμε για τις συνθήκες εργασίας, για την ποιότητα διαβίωσης και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Και έχουμε τρία ευρωπαϊκά παρατηρητήρια για τις συνθήκες εργασίας και έχουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις αλλαγές στη δίκηση και την αναδιάθρωση. Όπως είπε και ο Κρίστιαν, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη δραστηριότητα, παρόλο που θα πρέπει να περιμένουμε για το νέο προπολογισμό και να δούμε τι προσωπικό μπορούμε να έχουμε, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε αυτές τις βασικές δραστηριότητες στο μέλλον έλεγχος της ποιότητα των εργασιών και διεθνωτικές αλλαγές ε, λόγω της κρίσης είναι κάτι που μας απασχόλησε και πέρσι και φέτο. Παροχή πληροφοριών περί διαθρώσεων, αναδιαθρώσεων μέσω του παρατηρητήριου για την αδιάθρωση πάνω από 400 μέτρα υποστήριξης δημοσίευσαν στο σελίδα που εφαρμόζουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι κυβερνήσεις είδαμε ποιε είναι οι διαθωτικές αλλαγές στην αγορά εργασία. Η ύφεση επιτάχυνε τις διαθωτικές αλλαγές. Βασική τάση, η αγορά εργασία, οι αγορέ εργασία εξακολουθούν να απολώνονται. Ακόμα και κατά τη διάρκεια τη ύφεση δημιουργήθηκαν θέσει απασχόληση στην Ευρώπη, αλλά στα δύο άκρα. Με πολύ υψηλέ αμοιβέ και πολύ χαμηλέ αμοιβέ. Αυτά τα δύο επίπεδα. Αυτή είναι η γενική τάση. Σε κάποια κράτη-μέλη είδαμε διαφορετικέ εξελίξεις και έχει δημοσιευθεί μια έκθεση και είναι πλήρες κεφάλαιο στη βασική έκθεση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Ευρώπη 2011. Η των εργασιών εμπεριέχει πολλά στοιχεία. Και η έρευνα της συνθήκης εργασίας δείχνει πώς αλλάζουν στην Ευρώπη οι συνθήκες κατά διάρκεια 20 αιτίας. Συνεχίζεται η ανάλυση. Θα ξεκινήσει ενδελεχής ε, ε, έρευνα για την ποιότητα των εργασίων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Θα ξεκινήσουμε με δευτερεύουσες αναλύσεις και τόμε ε, οργανώσεις, τρόποι εργασίας και να βρούμε νέες προσεγγίσεις ανταγωνιστικές με στόχο καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και θα πάμε μετά στη νέα έρευνα για τις εταιρείες στην Ευρώπη και ποιες πρακτικές ακολουθούν το 2012 και το 2013 και άλλη ανάλυση των συνθήκων εργασίας θα εστιάζεται επί της γυράνσος του εργατικού δυναμικού, δεν θα σε εκπλήσει, διότι είναι το ευρωπαϊκό έτος για την ενεργοποίηση των ε, ηλικιωμένων εργαζομένων και στη Δανέζικη Προεδρία κάναμε μία από τις ε, ε, βασικές ε, παρεμβάσεις στο γεύμα παρέθεσε η Δανέζικη Προεδρία για το έτος. Ε, οι σχέσεις των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια της ανάκαμψης. Και μετά αμοιβέ μηχανισμοί ε, τα τιμαριθμικής προσαρμογής ήταν πράγματα που ενερευνήσαμε ε, σε σχέση με όλα αυτά που παρανέφερα. Αυτοί που επλήγησαν περισσότερο ήταν οι νέοι από την κρίση. Και ο φορέας μας, μαζί με τις άλλες τρεις, που είναι παρόντες έκαναν κοινό σεμινάριο στο Κοινοβούλιο. Θέλαμε να δείξουμε τη συμπληρωματική συνεισφορά των τριών υπηρεσιών μας. Έχουμε πρόγραμμα για τους νέους, τις ανάγκες που έχουν και εκτιμήσαμε το κόστος των αναγκών για 21 χώρες είναι 100 δις ευρώ το χρόνο. Και αυτή είναι η συντηρητική υπολογισμή. μπορούμε να κάνουμε μεγάλες οικονομίες. Μέχρι 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει κοινωνικό κόστος όμως. Δεν θέλουμε απομάκρυνση της συμμετοχής από την κοινωνία. Είδαμε άλλα στοιχεία που αφορούν αυτό το θέμα όσον αφορά την ποιότητα της διαβίωσης και την ποιότητα της κοινωνίας. Κάναμε συγκρίσεις αποτελεσμάτων και ερωτήσεις που απαντήθηκαν στο ευρωμανόμετρο. and we are currently finishing the field work of the third European Quality of Life Survey, so we will... Και τελειώνουμε και την τρίτη έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη και θα δημοσιεύσουμε φρέσκα απορίσματα φέτος. Με σχετικές πληροφορίες. Η ποιότητα ζωής λοιπόν. Προβλήματα πολιτών. Ετοιμάσαμε διάφορες εκθέσεις, κάναμε διάφορες έρευνες. Πώς γίνεται ο χειρισμός των χρεών των οικοκυριών καινοτόμε λύσει για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Επόμενος στόχο. για το επόμενο τετραετέ πρόγραμμα. Θα συζητήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτά τα θέματα. Ποια? Αντιμετώπιση της κρίσης και συνεκτική ανάκαμψη. Με αυτό θα ασχοληθούμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ η κυρία Μαντλέν Σερμπάν, το Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης, τελευταία παρέμβαση. Κάθε φορά πρέπει να λέω τις ιδιότητές σας και που, από πού είσαστε για να μην συγχαίω με τις έδρες. Είσαστε το Ίδρυμα του ε, Τωρίνου λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω ευχαριστώντας σας και εσάς και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας διότι το 11 μας βοηθήσατε πολύ. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και όπως και οι άλλοι συνάδελφοι θέλω και εγώ να ελπίσω ότι θα συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία και το 12 ίσως ακόμη και μετά. Ήρθα λοιπόν να σας εκθέσω τα πεπραγμένα μας του 11 Έχουμε μοιράσει και το έγγραφο και με την άδειά σας εγώ θα περιοριστώ τώρα σε τρία-τέσσερα στοιχεία από αυτά που αναφέρει. Θα πω μερικά λόγια για τις προτεραιότητες μας το 12. Όπως γνωρίζουν όλοι, το Ίδρυμα του Τουρίνου εργάζεται εξ ονόματος της Ένωσης για την εξωτερική διάσταση των προγραμμάτων της στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασυχόλησης. Το 11 λοιπόν είχαμε 30 εταιρικές συμφωνίες με τρίτες χώρες με βάση πάντα την εντολή που εσείς αποφασίσατε να μας χορηγήσετε σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Συμβουλεύουμε τις χώρες αυτές σε συνεργασία και με την Κομισιόν στους τομείς αυτούς και για να βελτιωθούν οι δυνατότητες τους για την καλύτερη διάδοση της γνώσης μεταξύ τους και, με, και διεθνώς, με τις διεθνείς οργανώσεις. Επειδή λοιπόν είμαστε έτσι σύμβουλοι, θα ήθελα να πω ότι πρέπει πρώτα να μιλήσω για τη διαδικασία του Τουρίνου. Η διαδικασία αυτή εμπνέεται από μια νέα εξέλιξη, δηλαδή μια άλλη διαδικασία, τη λεγόμενη της Κοπενχάγης, που μας την ανέφερε ο εκπρόσωπος του Σεντεφόπ. Είναι πολύ σημαντικό σε όλες αυτές τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε να βασιζόμαστε σε πραγματικά στοιχεία, όχι αυθαίρετα, όχι ad hoc και είναι επίσης σημαντικό η διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων αυτών να ε, περιέχει και ένα στοιχείο συμμετοχής των ενδιαφερομένων με εγγυημένη ποιότητα. Αυτά που σας λέω τώρα βασίζονται στην έννοια της καλής διακυβερνήσεως, good governance. Όταν συνάπτουμε συμφωνίες με αυτές τις χώρες θέλουμε να διασφαλίζουμε την καλή διακυβέρνηση, ότι μπορεί να επιτευχθεί δηλαδή καλή διακυβέρνηση. Και έτσι προσπαθούμε να, αυτές τις δυνατότητες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και σε αυτές. Φέτος συμπεριλαμβάνουμε ρητά αυτήν την ε, διάσταση της governance. Πώς όμως επηρεάζει η εργασία μας τις εξελίξεις στις χώρες αυτές, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Στη Μολδόβα το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία βασίζεται στη δουλειά μας, στη δική μας ανάλυση. Στο κοτσιφοπέδιο έχει εγκριθεί ένα στρατηγικό σχέδιο 11 με 16 για την παιδεία που πάλι βασίζεται σε δική μας ανάλυση με βάση τη διαδικασία του Τουρίνου στην Τινησία. Είχαμε την ευκαιρία να επιτηρήσουμε τον οδικό χάρτη απασχόλησης για να δώσουμε παραδείγματα. Στο Τατζικιστάν η ανάλυση μας κατέληξε στην έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας μιας νέας εργασιακής στρατηγικής. Αυτά είναι λίγα από τα παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω. Όλες αυτές οι χώρες επέδειξαν μεγάλο πνεύμα συνεργασίας και θεώρησαν, συμφώνησαν ότι η απασχόληση και η καταπολέμηση της ανεργίας είναι η τεράστια προτεραιότητα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Η Ουγγρική και Πολωνική προεδρία, προεδρίες το 2011 θέλησαν να παρουσιάσουν, είχα την καλοσύνη να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας μας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο η δουλειά μας γίνεται πιο δομημένη και έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα, δίνεται, της δίνεται μεγαλύτερη σημασία και στις χώρες μέλη. Με την άδειά σας λοιπόν, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο πλαίσιο προσόντων, στο προσοντικό πλαίσιο. είναι μια έννοια που προέρχεται, προκύπτει από αυτά που μας είπε ο συνάδελφος του Σεντεφόπ. Με μεγάλη χαρά λοιπόν μπορώ να σας πω ότι συνδιοργανώσαμε μια διάσκεψη με 67 χώρες, ξεπεράσαμε όντως τα σύνορα και τα όρια που μας είχαν τεθεί προηγουμένως. Η Ευρώπη εμπνέει και άλλες χώρες βλέπετε. Η εξωτερική λοιπόν διάσταση της δουλειάς μας θα, εξεταστεί, θα συνεχιστεί και το 12 γιατί η UNESCO θα οργανώσει το τρίτο της συνέδριο και μας εμπιστεύτηκε τη διοργάνωση της Ολομελίας για το θέμα των προσόντων και με μεγάλη χαρά θα φέρουμε στα μάτια του κόσμου ολόκληρου τη φωνή της Ευρώπης και τα επιτεύγματά της καθώς και τις δυνατότητές της συνεργασίας με αυτές τις χώρες. Πολλές χώρες λένε ότι γνωρίζουν εξελίξεις όπως στην Ευρώπη με πολύ ενθουσιασμό αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για να διασφαλίσουμε ότι τα κάνουν όλα όπως πρέπει και με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελούνται οι πολίτες και όχι μόνο στα χαρτιά. Δεν έχουν τελειώσει λοιπόν οι προσπάθειές μας, πρέπει να τις συνεχίσουμε και το 12. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας γίνεται για να διασφαλιστεί αυτό, ότι όλα τα προγράμματα εφαρμόζονται προς όφελος των πολιτών. Και στο νότο της Μεσογείου η Αραβική Άνοιξη μας έδωσε, μας έδειξε πολλούς καινούριου τρόπους συνεργασίας και συμβολής εν γέρος υποστήριξης των χωρών αυτών. Και είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε εδώ να σας αναφέρουμε ότι και η Τινησία και η Αίγυπτος επωφελήθηκαν από μας στον τομέα της παιδείας και της απασχόλησης. Δυστυχώς όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά το 12 στις 8 Μαρτίου θα αρχίσει, θα οργανώσουμε ένα πολύ συμβομαντικό συμβάν στην Τινησία με πρόσκληση της ΕΤΕ θα οργανώσουμε σεμινάρια απόκτησης προσόντων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τη σημασία που έχει ο νότος της Μεσογείου. Γιατί το 12 είναι το έτος γυράνσεως του πληθυσμού στην Ευρώπη, ενεργού γυράνσεως και πρέπει να δημιουργηθούν 60 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα σε 15 χρόνια. Εδώ η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει πολύ και η δική μας οργάνωση νομίζουμε ότι μπορεί να το κάνει. Ελπίζουμε να μπορέσει να το κάνει. Επίσης σημαντικό είναι τι συμβαίνει και στην Ανατολική Ευρώπη και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας αναλύοντας την σύνδεση προσόντων με απασχόληση στην Ουκρανία και στη Μολδόβα και θα προσπαθήσουμε να υποβοηθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη γιατί αλλιώς γιατί μάλλον είναι εξίσου σημαντικό να μιλήσουμε και για τα πράσινα προσόντα που δεν έχουν σύνορα, προσόντα δίχως σύνορα. Μιλάω για το 12, αλλά θέλω επίσης να προσέξετε τι κάνουμε και για τη μετανάστευση. Οι εταιρικέ σχέσεις για την κινητικότητα που έχουν συναυθεί με τη Μορδόβα αλλά και με την Αρμενία και με τη Γεωργία καθώς και με το Μαρόκο και την Τινησία είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι χάρη σε μας η εταιρική σχέση κινητικότητας με τη Μολδόβα τώρα συμπεριλαμβάνει και τα προσόντα και αυτό θα επεκταθεί και σε όλες τις άλλες τέτοιες εταιρικές σχέσεις. Τώρα γίνονται μελέτες για την προσοντική διάσταση της μετανάστευσης για να δούμε δηλαδή τι ακριβώς προσόντα έχουν και πρέπει να έχουν οι μετανάστες στην Ευρώπη και μία πρώτη μας, ένα πρώτο μας συμπέρασμα είναι ότι δυστυχώς οι πιο ειδικευμένοι και προσοντούχοι μετανάστες δεν απευθύνονται κυρίως στην Ευρώπη. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε καμία σχετική πρόταση σε όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε η συνοχή και η ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία είναι το κλειδί. Και το 12 λοιπόν αυτό θα τονίσουμε την εδαφική συνοχή στις χώρες με τις οποίες θα συνεργαστούμε. Τώρα για τη διαχείριση του προϋπολογισμού μας 97% των προβλέψεων χρησιμοποιήθηκαν και αυτό μας επέτρεψε να κάνουμε ό,τι κάναμε. Το 13 προβλέπονται περικοπές του προσωπικού και του προϋπολογισμού γιατί θέλουμε και οι ίδιες αυτές οι χώρες να αρχίσουν να δουλεύουν και όχι μόνο εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, μας εμπνέει ο ενθουσιασμός σας που σας έκανε να ξεπεράσετε και το χρόνο σας. Η κυρία και μετά ο κύριος φέρκας Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους καλεσμένους μας που ήρθαν για να μας δώσουν μία ενημέρωση σε σχέση με τις δραστηριότητες των φορέων τους. Χρειαζόμαστε αυτούς τους φορείς, δεν είναι μια πολυτέλεια η ύπαρξη των αποκεντρωμένων φορών, γιατί είναι φορείς οι οποίοι μπορούν να μας διαφωτίσουν καλύτερα για αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στο Ινστιτούτο του Μπιλμπάου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργαζόμαστε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ή μη δημοφιλές αν θέλετε, που είναι ακριβώς η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων που υπόκεινται σε την επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Θα θέλαμε να έχουμε την υποστήριξή σας στην εργασία μας. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο δεν δώσατε θετική απάντηση στην αίτησή μου να έχουμε την αρρωγή σας στα θέματα αυτά. Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό και το οποίο το έθιξαν πολλοί από τους σημερινούς ομιλητές, είναι η εξέλιξη των πλαισίων πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι νέες λοιπόν τα νέα προσόντα τα οποία χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης, όπως το τονίσατε και εσείς, η σύνδεση μεταξύ της μετανάστευσης, της εσωτερικής μετανάστευσης και των προσόντων. Αυτό είναι μια οπτική γωνία για την οποία θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις από εσά, γιατί εμείς εργαζόμαστε και στα θέματα της μετανάστευσης, της ενιαίας άδεια, της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη μέσα στις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές. Επίσης, όμως, θέλουμε να ξέρουμε για τα θέματα της εξέλιξης των προσόντων. Θα θέλαμε να έχουμε τα φώτα των αναλύσεών σας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να, έχετε, να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριος Θέρκας και η κυρία Μπάουερ μετά. Θέρκας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους διευθυντές και τις διευθύντριες των αποκεντρωμένων φορέων και εγώ υπογραμμίζω αυτά που είπε η κυρία Μωράν Σερτιέ σε σχέση με την αξιολόγηση που έχουμε για την προστεθέμενη αξία που αντιπροσωπεύεται στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και σε σχέση με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας μαζί σας. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις προφορικές παρουσιάσεις σας και για όλη την έγγραφη τεκμηρίωση που μας έχετε δώσει και που ίσως αναφέρεται σε ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι έχουμε τώρα στη διάστηση μας για να αναλύσουμε τα θέματα αυτά. Κάποια ερωτήματα. Καταρχήν ένα γενικό ερώτημα προς όλους σας. με λιγάκι από τα αποτελέσματα των δικτών που έχουμε δει. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου βασιζόμαστε σε κριτήρια αποτελεσματικότητας θα μας επιβάλλουν η κρίση και η λιτότητα του προϋπολογισμού να είμαστε πιο προσεκτικοί για τα θέματα αποδοτικότητας των φορέων αυτών. Επομένως, η σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτών και του κόστους κάθε φορέα θα γίνει πιο ανάγλυφη. Δεν ξέρω αν έχετε εκπονήσει τέτοιου είδου δείκτες, θα με ενδιαφέρε κάτι τέτοιο και αλλιώς θα ήθελα να σας αναφέρω ότι μια τέτοια απέτηση θα γίνει όλο και πιο έντονη τους επόμενους μήνες και χρόνια και για τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν πιο πολύ στην ομάδα μας, στην Επιτροπή μας, θα ήθελα να στραφώ στην Διευθύντρια του Ιδρύματος του Μπιλμπάου. Είχαμε προηγουμένως την επίσκεψη των ε, Υπουργών της Δανίας από την Προεδρία και έχουμε μείνει πολύ ανήσυχοι με κάποιες φήμες που κυκλοφορούν από την πλευρά της Κομισιόν που λέει ότι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται στον τομέα αυτό θα καθυστερήσουν και θα επιβραδυνθούν λόγω της κρίσης. Επρόκειτο όμως να γίνει μια συνδιάσκεψη για τα θέματα του λανσαρίσματος της νέας στρατηγικής. Μας είπαν οι δύο υπουργοί ότι κάνουν προσπάθειες για να διατηρηθεί αυτή η συνδιάσκεψη, αλλά υπάρχουν φήμες ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα είναι πραγματικά μια τραγωδία για την εκκίνηση αυτής της στρατηγικής. Αν εσείς τώρα μπορείτε να κάνετε και κάποια πρόταση επί τη βάση των δικών σας γνώσεων, για το πόσο σημαντικό είναι να γίνει η απαραίτητη αυτή επένδυση για να προχωρήσουμε στον δρόμο αυτό που αναφέρθηκε. Το δεύτερο ερώτημα πηγαίνει και αυτό στην ίδια κατεύθυνση. Έχουμε και πληροφορίες ότι η Κομισιόν θα ανακοινώσει μία σειρά κριτηρίων βάσει του στόχου της ε, μείωσης της γραφειοκρατίας και θα έχει σαν αποτέλεσμα να εξαιρέσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το κοινοτικό και εκτιμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πρόκειται για πάνω από 90% των ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη που χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική έχουν επωφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα και εδώ αν μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας και αν μπορείτε και εσείς να τονίσετε στην Κομισιόν ότι υπάρχει κάτι το οποίο ξεπερνάει τους οικονομικούς ισολογισμούς και είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το τελικό αποτέλεσμα, γιατί σίγουρα είναι καλύτερο να εργάζεται κανείς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουμε και την αστάθεια του εργατησιακού χώρου και τους κινδύνους. Για το, φορέα το, για το το φορέα της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να σας θέσω το εξής ε, ερώτημα. κάνετε μια πολύ σημαντική εργασία ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση να αναπτυχθεί περισσότερο στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι σε μια στιγμή που υπάρχει μια σημαντική μάζα εργαζομένων που πρέπει να αποκτήσει νέα προσόντα και δεξιότητες, θα ήθελα να ξέρω περισσότερο ποιες είναι οι έρευνες που κάνετε για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Στον κύριο Μέντες Βάλτης επίσης, του ιδρύματο του Δουβλίνου να σας θέσω δύο ερωτήματα τα οποία μα απασχολούν πάρα πολύ. Αναφερθήκατε στα δεδομένα της Eurostat για να καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η τάση των αναδιαρθώσεων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας πω, να σας ρωτήσω αν είσαστε διαθέσιμοι τη στιγμή που θα κάνουμε μία έκθεση στην Επιτροπή μας, αν είσαστε ε, έτοιμοι να δεχτείτε να ταξιδέψουμε στο Δουβλίνο, ο εισηγητής και οι σιώδες εισηγητές, για να δούμε ποια ακριβώς είναι η ανάλυση και η συμβολή σας στα φαινόμενα αυτά της αναδιάθρωσης, ώστε τα, με, τα, οι αναδιαθρώσεις αυτές να μην λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη, αλλά και όλες τις παραμέτρους. Επίσης, κύριε Βαλντές, αναφερθήκατε στον αντίκτυπο της κρίσης παρά στους νέους. Θα ήθελα να πείτε και κάτι πρόσθετο σε σχέση με τα θέματα αυτά. Και εν κατακλείδη. Στην κυρία Μαρτία Σερβάν, που είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε μαζί της στην επίσκεψη στο Τωρίνο, αν μπορεί να πει κάτι για τα προβλήματα υποδομών για τους ε, εργαζόμενους και τους ερευνητές στο Τωρίνο, αν έχουν βελτιωθεί αυτές οι συνθήκες. Αν, ή αν περιμένετε μονάχα από το Θεό και την Θεία Χάρη να βελτιωθούν τα πράγματα αυτά, ή κατά πόσον η κατα ποσο πράγματι προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές εφόσον τόσο σημαντική η εργασία σας. Υπάρχουν πολλές χώρες που ακολουθούν την διαδικασία του Τωρίνου. Συμβαίνει αυτό με όλες χώρες. Και επίσης, κυρία Ματλέν, τι γίνεται που τη στιγμή αυτή που υπάρχει μια νέα ευαισθησία. Πώς βλέπουν οι νέες αυτές κυβερνήσεις του αραγκού χώρου το θέμα της συνεργασίας μαζί σας και αν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνολική απόρριψη όλων των επιρροών από τον δυτικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπάουερ και μετά ο κύριος Πακ. Κυρία Μπάουερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις απευθυνόμενοι πρώτα προς τον εκπρόσωπο της ΟΕΣΑ της κυρίας Ρένατσεκ. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που υπάρχει το ΟΗΡΑ για την αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτό υπάρχει σε διάφορες γλωσσικές εκδοχές. Γιατί έτσι το μέσο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερη ερώτηση. Επισκεφθήκαμε το Ιδρυμά σας στο Μπιλμπάο και μας αναφέρθηκε τότε ότι παρά το ότι είναι παλιά υπηρεσία, δεν είναι κάτι καινούριο, παρόλα αυτά, δεν είχε συμφωνηθεί η διαδικασία καθορισμού έδρας. Ποια είναι η κατάσταση. Έχει επιτευχθεί συμφωνία. Και αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, τι μπορούμε να κάνουμε. Και για το Eurofund. Συμμετέχουν στην αξιολόγηση και αποτίμηση στρατηγικής για τους Ρωμά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπακ και η κυρία Μπεναρά του μετά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις τόσο ενδιαφέρουσες συνεισφορές τους και θέλω να θέσω καταρχήν ένα ερώτημα για το κοινωνικό σύστημα. Ξέρετε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις για άτομα ηλικιωμένα είναι εξαφάνιση για διάφορους λόγους. Αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το δίλημα και το δεύτερο ερώτημα το οποίο αφορά, ήθελα να τονίσω, είναι υπάρχει το ερώτημα του αν η ανεργία έχει διαρθωτικό χαρακτήρα Αν δηλαδή η Ευρώπη έχει μιζάρει υπερβολικά πολύ στον τομέα των τριτογενή της ε, παροχής υπηρεσιών ή αν η τρέχουσα κρίση στην απασχόληση είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Επίσης, σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση που έχουμε κάνει για τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας των τον τομέα εργασίας βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των ασθενειών, των ψυχικών ασθενειών που συνδέονται με το στρες. Επομένως είναι εργασιακά προκαλούμενες ασθένειες και συμπτώματα. Και φαίνεται ότι με την ε, αναθεώρηση της οδηγίας του 1999 για τις επαγγελματικές ασθένειες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό το στοιχείο και να βρεθεί μια λύση για τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Μπέναραμπάτου, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια και υγεία στον τόπο εργασία. Ποια ανάλυση για την υγεία των ανθρώπων εκτός των επιχειρήσεων ή των δομημένων οργανισμών μπορείτε να κάνετε. Αυτούς που εργάζονται, παραδείγματος χάρη, στο σπίτι τους. Οι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι. Τι ανάλυση κάνετε για την υγεία αυτών. Άλλη ερώτηση. Για τους μειοσκελετικά, μειοσκελετικά προβλήματα είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό για τι εταιρείε παραγωγή, αυτοκινητοβιομηχανία ή στα ταμεία, οι διοικητικέ θέσει. Όλε θέσει όπου υπάρχουν επαναλαμβανόμενε κινήσει. Άλλε ερωτήσει αφορούν το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την κατάρτιση του Τωρίνου. Πρώτο ερώτημα. Είπατε ότι δεν έρχονται εξειδικευμένοι μετανάστες στην Ευρώπη. Πού πάνε, στη ΣΥΠΑ, στην Κίνα, αλλού. Άλλο ερώτημα. Αναφερθήκα σημασία συνεργασίας με τις χώρες που υπήρξαν δημοκρατικές εξελίξεις, όπως Αίγυπτος, την Ισία. Η συνεργασία αυτή και σας ενδιαφέρει η κοινωνική προστασία, επεξεργαζόσατε το θέμα της κατάρτισης όσον αφορά τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνική προστασία. Ο κύριος Μπουλόν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω αυτούς που παρενέβησαν την ποιότητα των όσων είπαν και για τις δράσεις που ασκούν πέρα από τις δράσεις που αφορούν τον κάθε οργανισμό έχω κάποιος μια κάθετη, μια οριζόντια μάλλον ερώτηση που καλύπτει όλους. Απαντά όποιος μπορεί. Το ερώτημά μου αφορά τις κοινωνικές διαφορές. Διαφορές που υπάρχουν σε ολοκληρωμένη αγορά που προσπαθούν να ολοκληρώσουμε στο βαθμό του δυνατού. Διαφορέ που έχουμε σε κοινωνικό επίπεδο, υγεία, επαγγελματική κατάρτιση, συνθήκε εργασία κλπ. Δεν αναφέρω καν και του μισθού και τι συντάξει. Οι οργανισμοί αυτοί, στα πλαίσια των αποστολών του και των μέσων που χρησιμοποιούν, Ευρώπα, ΕΡΕΣ, Progress κλπ. Θεώρησαν ότι αυτές οι κοινωνικές διαφορές αποτελούσαν τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Εν τί αυτή περιπτώσει ανέλησαν την κατάσταση. Μπόρεσαν να, να αποτιμήσουν την κατάσταση, πρότειναν κάποια λύση, υπάρχουν κάποια εργαλεία που μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Ήθελα να το θέσω το πρωί αυτό το θέμα, το ερώτημα, όσον αφορά την κοινωνική σύγκληση στις ε, ε Δανές υπουργούς δεν το έθεσα το πρωί, το θέτω το ερώτημα τώρα, έμεσα. Στην Επιτροπή μας Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης έχουμε μία έκθεση που αφορά την καινοτομία και τις κοινωνικές, και αλλαγές. Συγγνώμη. Και ήθελε ο εισηγητής να κατευθυνθεί προς την κατεύθυνση της απασχόλησης. Όσον αφορά την έκθεση λοιπόν. Έχετε προτάσει όσον αφορά αυτό το πεδίο που καλύπτει η έκθεση καινοτομία και κοινωνικές αλλαγές στα πλαίσια τη βελτίωση της εργασίας. Και αυτό έχοντας υπόψη τι θέλουμε να πετύχουμε το στόχο της μεγαλύτερη κοινωνικής σύγκληση. Πρόεδρος. Να σας προτείνω να ξαναρχίσουμε με την ίδια σειρά. Διότι οι τέσσερις διευθυντής των αποκεντρωμένων υπηρεσιών δέχτηκαν ερωτήματα και ο καθένας θα απαντήσει στις ερωτήσεις που το ετέθησαν. Η κυρία Κρίστα Σέντλατσεκ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δεν ήταν κατά τη διάρκεια της θητείας μου που ετέθη αυτό το θέμα καλά. Αλλά ξέρω ότι πήραμε πολλές ερωτήσεις σε σχέση με τον αντίκτυπο, με το αποτέλεσμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία και την ασφάλεια. Αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε και ελπίζω ότι το έχουμε πράξει, αλλά φαίνεται ότι δεν σας έχει ικανοποιήσει, θέλετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το οποίο πράττουμε είναι να σας δώσουμε πληροφορίες σε σχέση με τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα τα στοιχεία αυτά της έρευνας για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια για να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Είμαστε στη χρονική φάση που ο φορέας μας θα πρέπει να δώσει να σας δώσει αυτά τα στοιχεία. Αυτό όμως το οποίο δεν κάνουμε και ενδεχομένω εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση γιατί όλα αυτά έλαβαν χώρα πρωτού αναλάβω εγώ ως, διευθυντής, ως διευθύντρια του Ιδρύματος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική αξιολόγηση. Δίνουμε στοιχεία, δίνουμε στοιχεία με τον πιο ουδέτερο δυνατό και αμερόληπτο τρόπο. Τα πρόσφατα στοιχεία, τα στοιχεία για όσες μετρήσεις έχουν γίνει και για τις πρακτικές λύσεις σε επίπεδο χώρου εργασίας. Δεν μπορούμε όμως υπό πολιτική έποψη να κρίνουμε τα θέματα αυτά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στα κράτη-μέλη. Εγώ έχω εργαστεί σε διάφορα κράτη-μέλη και τίθεται ένα θέμα ερμηνείας της ε, έρευνας. Είναι ένα πράγμα τα στοιχεία που προκύπτουν και ένα δεύτερο στοιχείο είναι η ερμηνεία αυτών των στοιχείων. Δεν είναι δικό μας καθήκον και δεν μας επιτρέπεται να αξιολογήσουμε εμείς από πολιτική άποψη τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την έρευνα για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αλλά φυσικά και εκεί έχουμε να κάνουμε ακόμα κάποιο έργο, μπορούμε να σας δώσουμε την πληροφορία που είναι διαθέσιμη και αυτό θα σας βοηθήσει να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις. Η δεύτερη ερώτηση που μου απευθύνθηκε αφορούσε το κατά πόσο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την εκπόνηση δικτών για, τους, για τις πολιτικές λιτότητος που επηρεάζουν το φορέα μας. Αυτό κατάλαβα, βεβαίως. Ένα από τα θετικά παραδείγματα είναι το δίκτυο των ε, αποκεντρωμένων φορέων. Συνεργαζόμαστε όλοι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το έργο των αποκεντρωμένων φορέων. Να σκεφτούμε παραδείγματος χάρη καλύτερα για ένα κοινό σύστημα κατάρτισης που μπορεί να παρέχεται σε όλους τους αποκεντρωμένους φορείς και έχουμε και άλλα σχέδια συνεργασίας για να μειωθεί το διοικητικό κόστος σε κάθε συγκεκριμένο φορέα. Η Ευρωπαϊκή Στατηγική για την Ασφάλεια αλλά και την Υγεία στην Εργασία από τότε που ξεκίνησα ως διευθύντρια στον φορέα του Μπιλμπάου ξεκίνησε η στρατηγική μας με το να πάμε χέρι-χέρι με την Κομισιόν και να ξεκινήσουμε μια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράλληλα με τις δικές μας ενέργειες. Συζητήσαμε με την Κομισιόν και νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία ότι θα ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο, θα υποστηρίξουμε στο βαθμό του δυνατού τη στρατηγική της Κομισιόν και η καταληκτική μου ημερομηνία για το φορέα του Μπιλμπάου είναι το τέλος του 2013. Αυτό συμφωνήσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά τη στιγμή που η Κομισιόν έχει αναβάλει τη δική τους καταληκτική ημερομηνία για τη στρατηγική τους, θα αναγκαστούμε και εμείς να προσαρμοστούμε στα δικά μας, να προσαρμόσουμε τα δικά μας χρονοδιαγράμματα με αυτά της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής αλλά υποστηρίζουμε πάντως και είναι πολύ σημαντικό σε καιρούς και οικονομικής πίεσης είναι απαραίτητο να έχουμε μια νέα στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας. Ένα περαιτέρω ερώτημα αφορούσε τον οικονομικό αντίκτυπο στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το 2012 ξεκινάμε τον προβληματισμό και τον αναστοχασμό μας για τον τρόπο που μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες για το πώς σε επίπεδο επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία, παραγωγικά στη διαδικασία αναδιάθρωσης μιας επιχείρησης, για να βελτιωθεί η κοινωνική πτυχή της αναδιάθρωσης χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, ακολουθώντας και το σχέδιο Κάιρης της Κομισιόν που έχει σαν στόχο να υπάρχει και μια κάπως πιο προληπτική μορφή αναδιάθρωσης των επιχειρήσεων. Επίσης, για την αξιολόγηση κινδύνων. <clears throat> Πράγματι, έχουμε ξεκινήσει τη μετάφραση του όηρα σε εννέα γλώσσες και μετά στις επόμενες σε μια επόμενη ομάδα γλωσσών στο βαθμό του δυνατού γιατί όπως είδατε με το όιρα είναι σχεδόν 17 κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν το όιρα και ενδιαφέρονται να πάρουν περισσότερα στοιχεία. Αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο, επομένω αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της εργασίας μας και χρειάζεται και να γίνει και η μετάφρασή του. Η συμφωνία ΣΥΤ μπορώ να, την, να σας ενημερώσω και να σας επικυρωσορίσω. Είχα μια πρώτη συζήτηση με, με την κυβέρνηση της χώρας των Βάσκων, ζητώντας να υπάρχει κάποια συμφωνία για τη συμφωνία ΣΥΤ. Ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση. Είναι πολύ σημαντικό ο φορέας του Μπιλμπάου να κάνει την εργασία του με τον σωστό τρόπο. Θα θέλανε να μας υποστηρίξουν, αλλά δεν μας δώσανε καμία συγκεκριμένη απάντηση σε σχέση με, χρηματική με χρηματοοικονομική υποστήριξη. Μας είπαν μπορεί ίσως να μας δώσουν ένα κτίριο στο Μπιλμπάου, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Και θα έχουμε και συζήτηση με τη νέα κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας στη Μαδρίτη, πάλι ζητώντας τους να μας δώσουν ε, υποστήριξη σε σχέση με τη συμφωνία για την έδρα μας. Είναι όλα αυτά υπό επεξεργασία οι γυράσκοντες εργαζόμενοι. Για να σας δώσω κάποιες ενδείξεις σχετικά. Ξεκινήσαμε πέρσι την ε, ανάπτυξη στοιχείων σε σχέση με τους γυράσκοντες εργαζομένους και το θέμα των ηλικιωμένων εργαζομένων σε επίπεδο επιχειρήσεων είναι από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν. Θα συνεχίσουμε την εργασία μας για να δούμε πώς μπορούν να προσαρμοστούν τα, οι χώροι εργασίας στις ανάγκες των ηλικιωμένων και πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τα εργαλεία τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική και ηλικιακή πολυμορφία και η έρευνα που έχουμε ξεκινήσει τώρα για την ηγετική θέση και την συμμετοχή θα συμπεριλαμβάνει και την πτυχή της πολυμορφίας του χώρου εργασίας σε επίπεδο επιχείρησης. Για τις ψυχοκοινωνικές κοινωνικές πτυχές της εργασίας, βέβαια πάντα αυτό είναι τμήμα της έρευνάς μας, η έρευνα αυτή έδειξε, κατέδειξε σαφώς ότι ο αντίκτυπος στην υγεία των εργαζομένων από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους αυξάνει σε όλους σχεδόν τους τομείς και εμείς αντιδρούμε ήδη στην εκστατεία μας για τις ηγετικές θέσεις και τη συμμετοχή. Ο στόχος μας είναι να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση από τη μία πλευρά, αλλά συγχρόνως από την άλλη πλευρά να δώσουμε λύσεις πολιτικές, στρατηγικές σε όλα τα επίπεδα και ξέρετε ότι το 2013 αλλά και το 2014 θα ξεκινήσουμε την εκστρατεία για τον ψυχοκοινωνικό κίνδυνο και προσπαθούμε μαζί με τους εταίρους μας να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα αυτό. Δεν γνωρίζω αν η τροποποίηση της οδηγίας του 1989 θα βοηθήσει πολύ, αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έλλειψη πληροφοριών, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό θέμα το να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση των εργαζομένων, αλλά είναι απαραίτητο να δώσουμε στις επιχειρήσεις και πρακτικά εργαλεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά σε συνεργασία με τα συνδικάτα και τους εργοδότες. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Ένα ακόμα ερώτημα που μου θέσατε ήταν ο εντίκτυπος της, στην υγεία των εργαζομένων που βρίσκονται στο σπίτι τους, που εργάζονται με τηλεργασία. Δεν είναι μέσα στην εντολή του φορέα μας. Παραδείγματο χάρη για την υγεία των γυναικών. Καλύπτουμε και την πτυχή των γυναικών που εργάζονται στην οικία τους. Και εκεί ο αντίκτυπο στην υγεία είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίκτυπο σε αυτούς που πηγαίνουν στο χώρο εργασίας που είναι κυρίως οι άνδρες. Έχουμε λοιπόν και εκεί ανάδραση για θέματα των ηλικιωμένων οι οποίοι αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό δεν είναι από τις ομάδες στόχου που αντιμετωπίζουμε. Εμείς κοιτάμε κυρίως τους εργαζομένους στις εταιρείε. Επίσης, έχουμε μια συνεχιζόμενη μελέτη για τις μειοσκελετικές διαταραχές γιατί αφορούν το, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων. Επομένως, έχουμε συμπεριλάβει στο σχέδιό μας για την ηλικία και μία δημοσίευση για τις διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος σε επίπεδο επιχειρήσεως που είναι και προέκταση του ε, προηγούμενου έργου μας και της εργασίας μας για το πώς να αποφύγει κανείς τέτοια προβλήματα υγείας και όπως ε, τονίσατε επομένω, ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η επαναληπτική εργασία και ο στόχος μας είναι να δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες πώς να αποφύγουμε τέτοιες αρνητικές συνθήκες στις εταιρείε. Δεν θέλω να σας ε, περικόψω, αλλά πρέπει να κλείσετε. Αυτά με ρωτήσατε, αυτά απάντησα. Μπορώ να δώσω το λόγο λοιπόν στον συνάδελφό μου τώρα, στον κύριο Λετ Προσπαθώ να είμαι σύντομος για τη μετανάστευση και τα προσόντα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε τη σωστή προσέγγιση. Όταν προσπαθούμε να πιστοποιήσουμε τα προσόντα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τους μετανάστες και να του βοηθούμε. Ξέρουμε ότι η αναντιστοιχία των προσόντων με την εργασία για τους μετανάστε είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επαλήθευση στην οποία προχωρούμε. Είναι πράγματι κομμάτι της εργασία μας, σημαντικό κομμάτι της εργασία μας. Θα υπάρξει ένα υπόμνημα στο τέλος του Φεβρουαρίου και μια ερευνητική έκθεση που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα των ερευνών μας, όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά η οποία εστιάζει και στα θέματα μετανάστευσης. Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, όπου δεν έχουμε ακόμα ικανοποιητικέ απαντήσεις, είναι το θέμα της γύρανσης. Και από τη μία μεριά έχουμε να κάνουμε με τις ανάγκες προσόντων για τους ηλικιωμένους, γιατί αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτά τα άτομα στην εργασία θα πρέπει να τους αναβαθμίσουμε, να επαναεπικυροποιήσουν τις, ε, τα προσόντα τους και συγχρόνως τα άτομα αυτά είναι αυτά που είναι πολύ πιο δύσκολο να τα προσεγγίσουμε και να τους αυξήσουμε τα προσόντα. Έχουμε μία σειρά από αρθρωτά τμήματα modules, γιατί είναι διαφορετικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αυτοί. Είναι θέμα που εμπλέκει την παιδαγωγία, εμπλέκει και τη χρηματοδότηση και έχει να κάνει με μια ειδική ομάδα που έχουν ανάγκη να μεταβούν σε άλλο πλαίσιο. Για τις εργασίες κατοίκων δεν είναι μονάχα το θέμα αυτό ένα θέμα που έχει να κάνει με την καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι ένα, μια κοινωνική τάση η οποία αναδύεται και θα έχει μεγάλη σημασία στο μέλλον. Και έχουμε κάνει σημαντική εργασία στο θέμα αυτό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο σπίτι και οι επιχειρηματίες που βρίσκονται στο σπίτι τους είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς απασχόλησης και πολλές από τις εργασίες του μέλλοντος θα έχουν αυτή τη μορφή. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να τύχουν κατάρτιση, να τύχει αναγνώρισης η κατάρτισή τους μέσα σε ένα πιο τυπικό σύστημα. Το προς το παρόν δεν βρίσκονται στο επίσημο σύστημα αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι ανισομέρεια. Όχι, δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα φυσικά είναι σημαντικό, αλλά μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης, αυτό το οποίο χρειάζεται να εξασφαλίσουμε είναι ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να τονίσουμε τη σημασία της ε, παιδείας για μια πιο ενεργό πολιτική ζωή και ζωή στην κοινωνία. Επίση, για τι δυνατότητε εξοικονομήσεω στου διάφορου αποκεντρωμένους φορεί υπάρχουν πάντα αυτέ τι δυνατότητε προσπαθούμε να τι αντιμετωπίσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Δύο παραδείγματα. Πέντε μέλη του ΣΕΔΕΦΟΠ, πέντε μέλη του προσωπικού του ΣΕΔΕΦΟΠ ήταν πέρσι μέρα και νύχτα σε αποστολέ. Οι αποστολέ είναι πολύ δάπανε, ιδίω όταν θέλει να πάει κανεί από Θεσσαλονίκη μακριά και εμείς διερευνούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις αποστολές αυτές. Δεύτερον, βλέπουμε αν μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις αποστολές σε βιντεοδιασκέψεις ή διασκέψεις μέσω Skype. Αυτά είναι παραδείγματα. Άλλα παραδείγματα φυσικά είναι ότι έχουμε προχωρήσει περισσότερο σε ηλεκτρονική δημοσίευση και επικοινωνία που είναι φθηνότερη από το χαρτί. Αλλά δεν θα ήθελα, θα να σας προειδοποιήσω ότι μια πολύ περιοριστική ερμηνεία για να επιτευχθούν εξοικονομήσεις θα περιορίσει και την αποτελεσματικότητά μας. Πολλές φορές έχουμε πολύ ε, ε, δύσκολα θέματα και γραφειοκρατικά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως είναι η προστασία δεδομένων που καταδαπανούν πολλούς πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα τα πω ισπανικά γιατί με βολεύει καλύτερα έτσι λοιπόν. Το πρώτο ερώτημα ήταν ένα γενικό ερώτημα για τους ενδείκτες. Αν έχουμε αποτελέσματα σε σχέση όχι μόνο με την αποτελεσματικότητα αλλά και την αποδοτικότητα. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς σε όλους τους προϋπολογισμούς που ισχύουν στην εποχή μας. Είναι πράγματι μια πραγματικότητα και σε όλους τους αποκεντρωμένους φορείς, τουλάχιστον στη δική μας. Ο προϋπολογισμός μας είναι 20 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε λιγότερα από 100 άτομα ε, στο οργανόγραμμά μας. Κατανοούμε λοιπόν τη σημασία αυτού του θέματος. Είναι υποδημοσίευση η έκθεση για το benchmarking που έχει εκπονηθεί από το Ελεκτικό Συνέδριο. Θα ήταν ενδιαφέρον όχι μόνο να συγκρίνονται μεταξύ τους οι επιχειρήσεις αλλά και με εθνικούς φορείς του ίδιου μεγέθους και διεθνείς φορείς ευρωπαϊκού επίπεδου που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή σύγκριση για μας. Εν πάση περιπτώσει, το 72% του προϋπολογισμού μας αφορά την έρευνα και την επικοινωνία, γιατί και αυτή είναι και η εντολή μας. Παράδειγμα, οι τρεις ευρωπαϊκές έρευνες που έχουν γίνει από τα τρία παρατηρητήρια καλύπτουν το 34% των πόρων μας. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας. Στη δεύτερη ερώτηση του κυρίου Θέρκας για τις αναδιαθρώσεις, η δραστηριότητά μας στο, ε, στο Ινδρυμά μας περιλαμβάνει και όλες τις πληροφορίες για την απώλεια και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σχέδια που έχουμε κάνει για την αναδιάρθρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμπληρώνουμε τώρα ένα σχέδιο που είναι η ανάλυση των διαδοτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και προφανώς, προφανώς θα μπορούσαν πάντα να γίνουν περισσότερο στα θέματα αυτά εφόσον έχουμε τους απαραίτητους πόρους. Το Ταμείο παγκοσμιοποίηση, παραδείγματο χάρη, είναι ένα χώρο όπου εμεί είμαστε σε πολύ καλή θέση να αξιολογήσουμε τα μέτρα αυτά ή επίση την παρακολούθηση θεμάτων συλλογικών απολύσεων και την πληροφόρηση για τις, ε, των εθνικών αρχών για τις συλλογικέ απολύσεις, το αν έχουν νομική ε, ε, αν έχουν νομική βάση ή όχι. Όλα αυτά τα δεδομένα μπορούμε πάντα να τα αξιολογήσουμε. Το σημαντικό πάντως είναι ότι είμαστε ίσως η πρώτη πηγή πληροφοριών για αυτά τα θέματα και γι' αυτό θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχτούμε μια επίσκεψή σας. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και πέρσι στην Επιτροπή Απασχόληση. Για την απασχόληση των νέων έχουμε δημοσιεύσει τα πρώτα αποτελέσματα και του χρόνου θα υπάρξει συνολική έκθεση όχι μόνο μια εκτίμηση του κόστους που αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και οι κοινωνικές επιπτώσεις και τα πολιτικά μέτρα τα οποία εφαρμόσουν τα κατι μελη οι κοινωνικοί εταίροι, ώστε να μπορέσει να προκύψει από όλα αυτά μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Για τα άλλα θέματα Όσον αφορά του ε, Ρωμά θα δημοσιεύσουμε, δεν έχει δημοσιευθεί ήδη στην ιστοσελίδα, δεν είμαι σίγουρο, ένα πρόγραμμα για τι συνθήκε διαβίωση αυτών που θα εστιάζεται στη στέγαση βασικά. Συγκεκριμένο αίτημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ λάβαμε αυτό το αίτημα και συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία της Βιέννης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι οργανισμός που φέρει τη βασική ευθύνη για αυτό το τομέα. για τους άλλους εργαζόμενους, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα στο Δουβλίνο, επί σειρά ετών, έκανε πολλή δουλειά για τη γύρανση του εργατικού δυναμικού και πώ μπορούμε να χειριστούμε το εργατικό δυναμικό. Έχουμε τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων πιθανότατα για τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο επιχειρήσεων για να διαχειριστούν το θέμα του γυράσκοντος εργατικού δυναμικού. Αυτό ε, ταιριάζει και με την εργασία που κάνουμε για τις συνθήκες εργασίας πρέπει να συμφιλώσουμε το έργο των ηλικιωμένων εργαζομένων που έχουν να φροντίσουν κάποιους ε, εξαρτώμενους ε, συγγενείς τους. Τώρα για την ανεργία. Αν είναι θεωτική ανεργία ή κυκλική. Φέτος, ήδη το 2012, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Δεν είναι εύκολο θα γίνει το παρατηρητήριο εργασιών. Στον οικοδομικό τομέα στην Ισπανία δεν θα καλυφθούν, δεν θα ξαναδημιουργηθούν οι θέσει που υπήρχαν πριν την κρίση. Αυτό είναι σαφέ. Είναι διθοτικό το πρόβλημα. Πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι άλλε δεξιότητες για να μπορέσουν να εργαστούν αλλού, σε άλλου τομεί. Σε άλλου τομεί δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η κατάσταση. Είναι τμήμα των εργασιών μα φέτο κοινωνικές διαφορές. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε συμπεριλαμβάνει την τάση που βλέπουμε από όλες εργασίες. Δηλαδή έχουμε ή εργασίες, θέσεις με πολύ υψηλές, υψηλές αμοιβέ ή με πολύ χαμηλές. Υπάρχει πόλωση. Και θέλουμε να δούμε ποιες πολιτικές λειτουργούν. Δεν είναι τα ίδια, η ίδια θελουμε να δουμε ποιες πολιτικες λειτουργουν δεν ειναι τα ιδια ιδια κατασταση σε όλες τις χώρες. Υπάρχει διαφορετική τάση στην αλλαγή του εργατικού δυναμικού. Και θα γίνει η τρίτη έκθεση για την ποιότητα διαβίωση στην Ευρώπη. Θα καλύψουμε περίπου 14 περίοδο. Θα δούμε ποιες είναι οι τάσεις. Πρόσβαση βασικές υπηρεσίες, παραδείγματο χάρη τι γίνεται. Βασικές συνθήκες διαβίωσης. Αυτά εξετάζουμε μεταξύ άλλων. Τα πρώτα πορίσματα της ε, έρευνας θα δημοσιευθούν φέτος και πιθανότατα του χρόνου προβλέπεται ότι η πιο διεξοδική ανάλυση ε, θα αφορά αυτούς τους συγκεκριμένους ε, τομείς και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε το κόστος των αποτελεσμάτων και ποια είναι τα κριτήρια επιδόσεων των υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μας ελέγχει, έκανε συστάσεις και πήρε υπόψη τις συστάσεις. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση ε, βρήκαν ότι είμαστε σε καλή θέση. Θα βελτιώσουμε την κατάσταση όμως, την αποδοτικότητά μας και πώς θα το πετύχουμε εξετάζουμε. Έχουμε ένα σύστημα που αφορά τη, τον χειρισμό της ποιότητας και της απόδοσης. Εξετάζουμε ε, πού μπορούμε να κάνουμε οικονομίες, σε ποιο τομέα. Και γι' αυτό μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο θα ξεκινήσουμε μια ανάλυση το Μάρτιο για το κόστος της διακυβερνήσεως του φορέα μας, Διοίκηση. Κάναμε πέρσι κάποια έρευνα όσον αφορά το κόστος των νεκρών. Στις εκθέσεις που σας υποβάλλουμε αναφερόμαστε στον αριθμό αποτελεσμάτων πρέπει να πετύχουμε με τα χρήματα που μας δίνεται. Σωστά είπατε όμως δεν, αρκεί, ε, η, δεν αρκούν τα ποσοτικά αποτελέσματα, χρειαζόμαστε και ποιότητα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα βήματα που κάνουμε. Υποδομές. Δεν έχω πολλά να σας πω. Δεν έχουμε ακόμα σύμβαση με τις Ιταλικές αρχές. Από αρχές Ιανουαρίου. Πολλές υποσχέσεις ακούμε. Παραμένουμε αισιόδοξοι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα μια σύμβαση και θα ξέρουμε πού θα συνεχιστούν οι εργασίες μας το 2012. Ο Επίτροπος, το γραφείο του Επιτρόπου μου ζήτησε ε, ενημέρωση. Η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακόμα μαζί μας. Την Παρασκευή θα έρθουν και μέλη, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε ότι έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα, στις χώρες της Νοτιού Μεσογείου μετά τις εκλογές και τις νέες κυβερνήσει που έχουν αυτέ οι χώρες. Πώς κινούμεθα εκεί. Κάθε νέα κυβέρνηση θέλει να διαφέρει την προηγούμενη. Αλλά δόξα τω Θεώ, η παιδεία, η απασχόληση και η κατάρτιση παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά. Διότι οι πολίτες είναι ακόμα στους δρόμους. Ψάχνουν για δουλειές. Ψάχνουν για κοινωνική και οικονομική προοπτική. Στην Τινησία έχει επιβεβαιωθεί ότι θα προχωρήσουμε. Στην Αίγυπτο διαφέρει πολύ κατάσταση. Μέσα Μαρτίου θα γίνει μια αποστολή εκεί. Δέχτηκε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Με ποιες οτερότητες δεν γνωρίζουμε. Είμαι σε στενή επαφή με την επιτόπου αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μαρόκο μετά τι εκλογέ Δεν άλλαξαν πολλά. σε ευθύνε στην κυβέρνηση και ρόλοι. Ο Βασιλιά ζήτησε νέα στρατηγική για την κατάρτιση και την παιδεία. Πε το ζήτησε. Και εκεί αυτό αποτελεί στοιχείο συνέχεια, Λιβύη. Το πρόγραμμα εργασιών το τροποποίησαμε, ξαποστάλαμε, αποστήλαμε και άλλαξε ξανά. Δεν είναι στο χαρτοκυφλάκι όμως ακόμα η Λιβύη. Μας ζητήθηκε όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσουμε εργασίες. Με το σύνθημα να κάνετε περισσότερα με λιγότερα. Μας είπαν άλλα χρήματα δεν έχει. Ψάχνουμε να βρούμε λύση. Ελπίζουμε ότι η Λιβύη θα εξακολουθεί να ωφελείται από ευρωπαϊκή στήριξη. Μετανάστευση. Ποιος είναι ο βασικός πρώτος προορισμός των μεταναστών. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις χώρες ανατολικής σα, Πάνε στη Ρωσία, νότια συνεργασία, πάνε στις χώρες του κόλπου. Και έχουμε άλλες πληροφορίες να σας δώσουμε. Μπορούμε να σας δώσουμε λεπτομέρειες αν θέλετε όσον αφορά τη μετανάστευση δεξιοτήτων. Το σημαντικό χρειάζεται δουλειά για, το, για την προσέλκυση ταλέντων. Η γερμανική κυβέρνηση μας ζήτησε να κινηθούμε όσον αφορά τους πιο ειδικευμένους ανθρώπους και θα κινηθούμε καταλήλως με κοινέ δράσεις. Κάνουμε πολλά για την προετοιμασία εξετάσεις του θέμα της μετανάστευσης. Ελπίζουμε ότι οι καλύτερες δεξιότητες από τούδε και στο εξή θα έρχονται στην Ευρώπη. Κοινωνικές διαφορές. Κάνουμε αναλύσεις. Και φέτος θα κάνουμε ανάλυση. Και θα δούμε αν οι χώρες εταίροι μας εξετάζουν την οικονομική και κοινωνική σύγκληση διότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές διαφορές στις χώρες. Στο έργο μας συμπεριλαμβάνουμε την κοινωνική προστασία. Αυτά και ευχαριστώ και ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς φτάνουμε στο τέρμα των, της συζήτησης αυτής που ήταν τόσο πολύτιμη. Δυστυχώς έτσι γίνεται πάντοτε. Θα έχουμε όμως και άλλες ευκαιρίες να ανταλλάξουμε απόψεις και χαίρομαι γι' αυτό ιδιαίτερα. Είτε γιατί εσείς θα αναλάβετε πρωτοβουλίες όπως τη διάσκεψη που οργανώσατε πέρυσι, είτε γιατί και αν κάνετε την πρωτοβουλία επαναλαμβάνω εμείς θα ανταποκριθούμε και τα λοιπά ε, ε, είτε γιατί θα έχουμε άλλες ευκαιρίες ως αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας να επισκεφθούμε φέτος το Ίδρυμα του Τουρίνου και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και για να είναι ισορροπημένα τα πράγματα θα αλλάξουμε τις προεδρίες. Εγώ θα προεδρεύω τις αποστολή στη Θεσσαλονίκη και άλλος θα προεδρεύει στο Τουρίνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία για το 2012. Ίσως πρέπει να δούμε με την Κομισιόν πώς μπορούμε ως Κοινοβούλιο να σας κινητοποιούμε πιο ενεργά, να σας καλούμε ανάλογα με τις ανάγκες μας. Πέρσι μιλήσαμε με μερικούς από εσά και όταν σκέφτομαι θέματα όπως την αξιολόγηση των μέτρων λιτότητας σε ορισμένες χώρες ή τους κινδύνους που εμπεριέχουν τα μερικά προγράμματα εκπαιδευτικά, αυτά είναι πολιτικά θέματα και χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη σας. Εκτός από την Κομισιόν λοιπόν θα μπορούσαμε να βλεπόμαστε και εμείς συχνότερα. Με βάση βέβαια τα προγράμματα που μας αναφέρατε, που μας δίνουν ήδη μία αντίληψη γενικότερα του τι μπορούμε να περιμένουμε. Τελειώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο και τώρα στο 19 δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Τσίμερ για να εξετάσει το σχέδιο γνωμοδότησή για την εφαρμογή τη αρχή τη ισότητα αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών με ογιαόμια εργασία ή εργασία τη αυτή αξία. Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή των Γυναικών όπου η εισηγήτρια είναι η Εδίθ Βάουερ και γνωρίζει καλά τα της δικής μας Επιτροπής. Ορίστε κυρία Τσίμερ μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σημείο αυτό της ημέρας διάταξης αφορά ένα θέμα το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, αλλά εξακολουθεί να είναι στον πυρήνα της εργασίας μας. Και πρέπει να τονίσω ότι από την εποχή που είχαμε συζητήσει για τελευταία φορά αυτό το θέμα και είχαμε καταλήξει σε μία άποψη σε μια θέση της Επιτροπής μας, δυστυχώς τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε και πάλι μια γρομοδοτηση για το θέμα αυτό. Η βασή, η για την ίση αμοιβή της ε, ίσης αμοιβής για ίση εργασία βρίσκεται ήδη στα άρθρα της συνθήκης και στις αρμόδιες οδηγίες Παρ' όλα αυτά, η ψαλίδα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών τα τελευταία χρόνια δεν έχει τροποποιηθεί. Στην πρόταση λοιπόν ρομοδότη μου, εγώ επικρίνω το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν υπήρξε κάποιο πρόγραμμα εργασίας μετά από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου το 2008, ούτε κάποια πρόταση για το 2012. Στα 27 κράτη-μέλη και τις, η, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξακολουθεί να υπάρχει μία διαφορά η οποία φτάνει Ε, ε, του επίπεδου 25% μεταξύ ανδρών και γυναικών και στη Γερμανία ακόμα και μεταξύ ατόμων με υψηλά προσόντα φτάνει το 23% αυτή η διαφορά. Βάσει των στοιχείων που έχουμε υπάρχει και διαφορά <coughs> στις συντάξεις 6 με 16% και 23% για αυτούς που βρίσκονται στο κατόφλι της ένδειας. Και επίσης η συμμετοχή των γυναικών είναι πολύ περιορισμένη στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί είναι τόσο μεγάλη η διαφορά αυτή στην αμοιβή ανδρών και γυναικών, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Μετά από διάφορες μελέτες, έχει φανεί ως τα δύο τρίτα των περιπτώσεων που υπάρχει μισθολογική ε, διαφορά, αυτό οφείλεται σε διάκριση λόγω φύλου. Και πράγματι, οι άνδρες που κάνουν την ίδια εργασία με τις γυναίκες κατατάσσονται σε υψηλότερη κλίμακα και επίσης υπάρχουν άλλες μορφές ε, διακρίσεων που θεωρείται πολλές φορές η ευελιξία πέραν των ορών εργασίας ως θετικό στοιχείο και είναι προφανές ότι οι γυναίκες που έχουν οικογένεια είναι λιγότερο ευέλικτες και επομένως έχουν χαμηλότερες αποδοχές. Οι γυναίκες εργάζονται στις λιγότερα αμοιβόμενες <clears throat> θέσεις εργασίας και επαγγέλματα και οι άνδρες στα υψηλότερα αμοιβόμενα επαγγέλματα. Υπάρχει λοιπόν μια, ένα μορφή διαχωρισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες που έχει ακριβώς αυτή την επίπτωση για την ψαλίδα των αποδοχών και επίσης οι γυναίκες έχουν λιγότερη συμμετοχή στις θέσεις ε, εξουσίας. Ο παραδοσιακός ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικογένεια είναι ότι αυτή είναι υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών και επομένως πλήττεται και από αυτό το στοιχείο. Είναι πολύ πιο συχνό η γυναίκα να διακόπτει για μεγάλο χρονικό διάστημα την εργασία της κτλ. Εμείς λοιπόν συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό ε, θα πρέπει να τονιστεί από τη δική μας πλευρά στη γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή Γυναικών και να συμπεριλάβουμε αυτές τις απόψεις στο ψήφισμά του. Εμείς στις ε, προτάσεις μας θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη να ληφθούν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να ξεπεραστούν τα στερεότυπα, ο διαχωρισμός ανδρών και γυναικών σε οριζόντιο και κάθε το επίπεδο, να ξεπεραστεί η μισθολογική διαφορά, να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι χρειάζονται και νέα στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να, μπορούν να, υπάρξει, να μπορεί να υπάρξει μια πιο συνεκτική σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών και να προσαρμοστούν αυτά στις νέες προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας δεν θα πρέπει να υπολογίζουμε μονάχα τις ε, ακαθάριστες αποδοχές ανά ώρα, αλλά και ένα σύνολο ενδεικτών, παραδείγματος χάρη την απόδοση μπόνους και πριν, γιατί και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Χρειαζόμαστε να έχουμε άμεσους συνομιλητές για τα μέτρα αυτά από την πλευρά της Κομισιόν και επίσης θα χρειαστεί να έχουμε και την άποψη των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων για να δούμε κατά πόσο υπάρχει κάποια δυνατότητα να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, αν μπορεί ήδη και σε πανεπιστήμια και όπου βρίσκονται τέτοια προβλήματα να υπάρξει μια μεγαλύτερη προσέγγιση και προφανώς εννοείται ότι πρέπει και με δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις να εξασφαλίσουμε ότι για ίση εργασία είναι ίση η αμοιβή. Δεν πρόκειται λοιπόν μονάχα για ένα πολιτικό ε, εγχείρημα πυθούς αλλά και για ένα νομικό εγχείρημα. Τώρα, η πρότασή μας περιλαμβάνει μέτρα ε, γενικά και ε, πολιτικές και επίσης νομοθετικά μέτρα. Καταρχήν την μεγαλύτερη χρήση του mainstreaming των φύλων για να ξεπεραστούν οι ανισορροπίες και οι ανισότητες να υπάρξει μια καλύτερη πολιτική για την ευελιξία στην εργασία, καλύτερη πολιτική για τη φροντίδα των παιδιών, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας συζήτησης που φυσικά είναι αντικείμενο τεράστια συζήτηση σε πολλά κράτη-μέλη και πιστεύω ότι κάτι ακόμα που θα ήταν χρήσιμο θα ήταν να έχουμε και κάποιο πιστοποιητικό ποιότητα των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. Υπάρχει επίσης και η συζήτηση η οποία έχει λάβει η χώρα για τις ποσοστώσεις σε σχέση με τις γυναίκες στις επιχειρήσεις. Έχει αυτό κάποιο νόημα για να μπορέσει να κλείσει κάπως η ψαλίδα αυτή. Η Νορβηγία αυτή τη στιγμή είναι η μόνη χώρα η οποία έχει υποστηρίξει μια, μια ε, επιβολή ποσοστώσεων στα διοικητικά συμβούλια για την ίση συμμετοχή των γυναικών και επομένως μπορούμε να λάβουμε την Νορβηγία, η οποία έχει καταφέρει να εξισώσει το ποσοστό άνδρων και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ως ένα παράδειγμα. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να συζητηθεί είναι ο βαθμός στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αποδεχθεί την έννοια της ε, ευέλικης ασφάλειας και να δει σε ποιο βαθμό η ευελιξιασφάλεια αυτή επηρεάζει το χάσμα στις αποδοχές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσον υπάρχουν θετικές επιπτώσεις της έννοιας της ευελιξιασφάλειας στο να ξεπεραστούν τα θέματα διακρίσεων. Αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα έρευνα για να την κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δω τώρα πώς τη λένε αυτή την κυρία. Σκυρσντέλφσκα. Και μετά η κυρία Εστρέαβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ καλά φέρατε το όνομά μου. Γιατί είναι και δύσκολο. Πρώτα πρώτα όμως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τσίμερ για την, για την τόσο ωραία γνωμοδότησή της. Η διαφορά μεταξύ μισθών ανδρών και γυναικών που κάνουν την ίδια εργασία ή την εργασία αυτής αξίας η διαφορά δεν μειώθηκε. Μερικοί μάλιστα λένε ότι οι κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν διαφορετικούς μισθούς δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί ότι είναι πιο χαμηλόμιστες οι γυναίκες είναι πια μέρος των κοινοτυπιών που ε, δέχονται όλοι. Θεωρείται ότι η δουλειά των γυναικών έχει λιγότερη αξία από των ανδρών και οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι πιο λιγότερο αποτελεσματικές, λιγότερο παραγωγικές. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαφή κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της αντρικής και γυναικείας εργασίας για να βασιστούμε σε γεγονότα και όχι σε ιδέες και προκαταλήψεις. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να ρωτήσω μάλλον, εάν είναι παρόν, να του ζητήσω να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της κοινωνικής μελέτης που έγινε από την Κομισιόν με στόχο να φανεί τι φρονούν οι επιχειρήσεις για αυτό το θέμα και αν έχουν συνείδηση ότι ασκούν άνηση μεταχείριση. Αλλά η έρευνα αυτή αφορούσε και το ευρύτερο κοινό με σκοπό να δείξει τι πρότυπα υπάρχουν και αν υπάρχει ισορροπημένη αντίληψη για τα δύο φύλλα. Για την κυρία Τσίμερ θα ήθελα να πω ότι η στρατηγική της ασφαλιξίας την οποία αναφέρει στη γνωμοδότησή της ως εργαλείο καταπολέμησης των ενισοτήτων αυτών σωστή, σωστή. Στο 6, στο σημείο 6, μιλάει για συνυπευθυνότητα. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι πρέπει και οι άντρες να, συμμετέχουν στα οικιακά και στη φροντίδα των παιδιών. Αλλά, αυτά να τα αποφασίσουν οι ίδιες οι οικογένειες, να, κατα... αποφασίσουν μόνες τους ποιο πρότυπο προτιμούν και να μην επιβάλλουμε εμείς την αλλαγή του συνήθους προτύπου κατανομής των εργασιών, καταμερισμού των εργασιών. Η κυρία Τσίμερ είναι υπέρ της παρακολούθησης και εποπτείας της εξέλιξης των μισθών και εγώ συμφωνώ γιατί δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια οι γυναίκες δεν ξέρουν πολλές φορές ότι οι άντρες συναδελφοί τους που δουλεύουν δίπλα τους πληρώνονται πολύ καλύτερα από εκείνες. Για την ίδια εννοείται. Έχουν αναλυφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες από κράτη-μέλη, τις ανέφερε η κυρία Τσίμερ και μόνο μία πανενοσιακή τέτοια έρευνα θα μπορούσε να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά τις ανισότητες αυτές στη μισθοδοσία άμα γίνει και μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε εδώ και τις οικογενειακές επιχειρήσεις όπου η ανισότητα των μισθών υπάρχει, υπάρχει ή καμιά φορά δεν υπάρχει καν μισθός για την σύζυγο. Καν. Πράγμα το οποίο έχει επιπτώσεις βέβαια για την σύνταξη ή μη σύνταξή της. Οι διαφορές των μισθών για την ίδια εργασία πρέπει να είναι η βάση και όχι οι προσφορές μισθών για αντρών που δεν κάνουν την ίδια εργασία με τις γυναίκες. Υπάρχει σχετικά μια πολύ καλή έκθεση της κυρίας Μπάουερ από το 8 και ελπίζω η Κομισιόν να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της τη χρονοδότησή μας. Ευχαριστώ. Εστρέλα Οβίρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγητρία. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό έργο. Η γνωμοδότηση αυτή καλύπτει ουσιώδη στοιχεία των εργασιακών σχέσεων και ιδίως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών συνδέεται άρρηκτα και με τη δυσκολία συμφιλήσεω της οικογένειακή με την επαγγελματική ζωή. Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τα στερεότυπα του φύλου, τα οποία διατρέχουν την κοινωνία μας. Και υπάρχουν φυσικά και αρνητικοί αντίκτυποι της ανισότητας αυτής των αμοιβών σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, αλλά ιδίως όταν φτάνουν οι γυναίκες στην σύνταξη. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτή η διαφορά αμοιβών ανδρών και γυναικών και τον τελευταίο καιρό αντίθετα με αυτό το οποίο είχε γίνει σε άλλους τομείς υπήρξαν υποχωρήσεις. Το 2005 η μέση διαφορά ήταν της τάξης του 15%. Αυτή τη στιγμή Τώρα έχει ξεπεράσει και το 17-18% κατά μέσο όρο. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου αυτή η διαφορά φτάνει μέχρι και το 30%. Επομένως έχουμε να αντιμετωπίσουμε de facto ένα σοβαρό πρόβλημα και το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκονται οι γυναίκες σε υποχρέωση να εργάζονται περισσότερο, περισσότερες μέρες το χρόνο, δύο μήνες το χρόνο περισσότερο κατά μέσον όρο, για να μπορέσουν να κερδίσουν τα ίδια λεφτά με τους άντρες. Το ένα έκτο δηλαδή του χρόνου παραπάνω. Ένα άλλο θέμα που συνάπτεται με τα θέματα της ανισότητας αυτής είναι και η μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Είναι απαράδεκτο από πλευράς κοινωνικής δικαιοσύνης και από πλευράς ισότητας μεταξύ των δύο φύλων να παραμένει αυτή η διαφορά αμοιβών και έχει προφανώς και οικονομικές επιπτώσεις αυτή η διαφορά. Γιατί το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι σχεδόν 10% μικρότερο από το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών. Εάν θέλουμε να λάβουμε υπόψη των στόχο της ε, στρατηγικής Ευρώπης 2020 να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας και να φτάσει το 70% είναι φανερό ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μονάχα με μία αύξηση σημαντική της απασχολησιμότητας των γυναικών. Επομένως, θα πρέπει να επιζητήσουμε την επίτευξη ισότητας τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανδρών και γυναικών, <clears throat> γιατί αυτό θα μας οδηγούσε σε αύξηση κατά 20 εκατομμύρια στον αριθμό των εργαζομένων. Αυτό θα έχει θετικέ συνέπειε για την οικονομία, γιατί βάσει των μελετών που έχουν γίνει, υπολογίζεται ότι η ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας θα είχε και αποτέλεσμα την αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 4 με 8% αν φτάσουμε αυτό τον αριθμό των 20 εκατομμύριων προσθέτων εργαζομένων μεταξύ των γυναικών. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δεχόμαστε αυτή την διάκριση η οποία υπάρχει και η οποία είναι αρνητική από κάθε άποψη και επίσης θέλω να προσθέσω το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες εργάζονται πολύ πιο συχνά σε επισφαλείς θέσεις εργασίας και σε εργασίες μερικής απασχόλησης. Περίπου 30% όλων των γυναικών κάνουν εργασία μερικής απασχόλησης, ενώ είναι μόνο 7% το ποσοστό αυτό για τους άνδρες που εργάζονται με μερική απασχόληση. Όπως ε, τόνισα, όλα αυτά έχουν αρνητική επίπτωση στην ε, συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και επίσης έχει καταδειχθεί ότι αυξάνει η διαφορά σε αποδοχές όταν οι γυναίκες όταν πρόκειται για πιο υψηλά αμοιβόμενες εργασίες. Επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες που είναι σε φάση μητρότητος, όπου θα πρέπει να λαμβάνεται αυτό υπόψη και να, να λαμβάνουν τις πλήρες αποδοχές τους κατά την περίοδο αυτό. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στις προτεραιότητες της ε, Δανικής Προεδρίας, οι οποίες και αυτές ακολουθούν την κατεύθυνση που διαγράφει η γνωμοδότηση αυτή της κυρίας Τσίμερ και που υποστηρίζονται και από την ομάδα των σοσιαλιστών ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και πιο συγκεκριμένα στον οικονομικό στίβο. Και όπως είναι γνωστό, υπάρχουν μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι μόνο 5% είναι το επίπεδο της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης απόφασης σε υψηλά επίπεδα των επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό αν σκεφτούμε ότι στο υψηλό αυτό επίπεδο δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα η οποία να είναι παραγματικά χάρη επικεφαλής μιας κεντρικής τράπεζας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Κομισιόν είχε προτείνει ότι θα παρουσίαζε στην αρχή του έτους μία πρωτοβουλία νομοθετικού χαρακτήρα για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια των δημοσίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα πάρει αυτά τα μέτρα <clears throat> που είναι απαραίτητα για να εξαλειφθεί αυτή η μισθολογική διαφορά ανδρών και γυναικών και να δοθεί ένας πιο σημαντικός ρόλος στις γυναίκες και στον οικονομικό στίβο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Madame Ovir, puis Madame Bauer. Κυρία Ovir και μετά Bauer. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τσίμερ και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα πρόβλημα. Η διαφορά στην αμοιβή υπάρχει και σε οριζόντιο επίπεδο. Υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη κάποια, κάποια επαγγελματική κλάδη που είναι ουσιαστικά κλειστή και είναι μόνο για τους άνδρες, οι οποίοι κερδίζουν περισσότερα χρήματα και επομένως συμβάλλουν στην ψαλίδα αμοιβών. Οι στατιστικές μας καταδεικνύουν ότι, ότι ακόμα και το ότι το 2007 μάλλον ήταν 7,5% η διαφορά αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως που βρισκόμαστε στην οικονομική κρίση, τα πράγματα πιστεύω ότι είναι χειρότερα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα 17 και όχι 7%, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει καμία μελέτη παρά το γεγονό ότι η κυρία Μπάουερ το 2008 στην έκθεσή της το είχε ζητήσει. Πέρσι στην πατρίδα μου στην Εστονία είχε αυξηθεί από 13% σε 38% η διαφορά αυτή. Η τάση αυτή λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας τρομάζει. Μπορούμε να συντάξουμε και να εγκρίνουμε εκθέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο μέτρο στο πλωστάσιό μας για να πείσουμε τις κυβερνήσεις να πράξουν κάτι. Γι' αυτό, ίσως ακριβώς το λόγο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα του προβλήματος αυτού. Θα πρέπει να ζητήσουμε νέες στατιστικές. Δεν έχουμε νέα στοιχεία με το 2007 και σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχουν καν νομικές ρυθμίσεις που να απαιτούν ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών για ίση εργασία. Γιατί το λέω αυτό. Στην Εστονία ενεκρίθη βέβαια η νομοθεσία κατά των διακρίσεων και στην νομοθεσία αυτή απαιτεί το να υπάρξει μια εξίσωση των αμοιβών για ίση εργασία. Ενεκρίθη αυτή η νομοθεσία το 2008, έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα οι οργανώσεις των γυναικών έχουν ζητήσει να εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο νόμος, αλλά στην πραγματικότητα νίξ. Και βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήμασταν στην προηγούμενη, στον προηγούμενο αιώνα. Επομένως, θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποτε η ρήτρα των συνδικών ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών. Ακόμα ένα πρόβλημα έχω να σας επισημάνω. Σας είπα ότι έχουμε μονάχα οριζόντιους δείκτες. Το, η ψαλίδα αμοιβών υπάρχει επίσης γιατί δεν ξέρουμε πολύ καλά και πόσο ψηλές είναι οι αποδοχές. Σε πολλά κράτη-μέλη είναι απόρριτες οι αποδοχές των εργαζομένων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες δεν ξέρουν ότι παίρνουν για την ίδια εργασία λιγότερα λεφτά από τους άνδρες. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει κάποια ενέργεια για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν όλοι μας με την Επιτροπή Γυναικών για να επιστήσουμε καλύτερα την προσοχή τους στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπάουερ και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κύριο Στάιν είναι παρόν και του απευθύνθηκε άμεσα ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Μπάουερ. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την γνωμοδότηση. Θεωρώ ότι είναι περιπλοκότατο ζήτημα. το να επανερχόμαστε στο θέμα αυτό μετά το 2008 είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Διότι έχει αλλάξει εντελώ η νομοθεσία. Γνωρίζουμε ότι είναι το παλαιότερο κομμάτι της νομοθεσίας όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Από τη συνθήκη της Ρώμης προέρχεται, του 1957. Βασικό μου ερώτημα που με απασχολούσε και όταν έγραψα και την προηγούμενη έκθεση επί του θέματος είναι το εξής. Πώς έχουμε νομοθεσία δευτερογενή 30 ετών χωρίς σχεδόν να έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημά μας που πρέπει να μας απασχολεί ως νομοθέτες. Τι να κάνουμε από αυτούς τους όρους. Να περιμένουμε και να κάνουμε πάντα εκστατείς ευαισθητοποίησης. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το εκτιμώ. Το μόνο θετικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την έκθεση του 2008 ήταν που ξεκίνησε την ημέρα για την ίση e αμοιβή. E Πολύ ενδιαφέρον βήμα, σημαντικότατο, όμως Γνωρίζουμε ότι η οδηγία για την αναδιατύπωση που αντικαθιστά την παλιά οδηγία για την ε, ισότητα στην πράξη δεν συνεπέφερε νέα μέτρα και σημαντικές αλλαγές. Βασικό μου ερώτημα είναι τι να κάνουμε υπ' αυτές τις συνθήκες. Να παραμείνει αυτή η νομοθεσία χωρίς κυρώσεις, χωρίς σαφή αιτήματα για διαφάνεια και να πιέζουμε τις διάφορες χώρες για να κάνουν πιο διαφανή τα συστήματά τους. Να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε ξανά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει νέα νομοθεσία. Προβλεπόταν πριν την προετοιμασία του οδικού χάρτη. Θα θυμόσαστε ίσως ότι πριν από δύο χρόνια είχαμε έναν οδικό χάρτη. Περίπου πριν από δύο χρόνια. Μα τον είχε στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χάρτης αφορούσε την ισότητα των φύλων. Τότε δεν έγινε αποδεκτός. Ερώτημα. Τι να κάνουμε τώρα υπό αυτές τις συνθήκες. αν ακολουθήσουμε τον δρόμο που επελέγει το 2008 και ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει βελτιωμένη νομοθεσία το 2013 ή αν ακολουθήσουμε κάποιες συγκεκριμένες προσεγγίσεις στον κοινωνικό διάλογο ή τέλος πάντων κάτι παρεμφερές Τελικό σχόλιο. Στα πρόσφατα στοιχεία του Eurostat, στην ιστοσελίδα είδαμε ότι ενημερώθηκαν τα στοιχεία. Όσον αφορά τη διαφορά των αμοιβών με βάση το φύλλο. 17,1 ήταν το στοιχείο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν στοιχεία που μιλούν από μόνο τους. να δώσω τον λόγο στον κύριο Ανδρέα Στάιν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει βασικά στο ερώτημα τη κυρία Σκουτζευνιέσκα. Σκουτζνιεύσκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορώ να πω ότι συμφωνεί απόλυτα με το βασικό πνεύμα της συζήτησης και με το σχέδιο γνωμοδοτήσεως ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά των αμοιβών με βάση το φύλλο ανδρών και γυναικών. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ισότητα των αμοιβών την έκανε μία από τις προτεραιότητες στα πλαίσια της στρατηγικής ισότητα ανδρών και γυναικών περίοδος 2010-2015. Στα πλαίσια της λόγω στρατηγικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε διάφορες ανακοινώσει. Αφορούσαν τα βήματα που θα εφάρμοζε για την εκτέλεση στρατηγική και θα προσπαθούσε να βελτιώσει την κατάσταση αφορά τη διαφορά μη ανδρών και γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφήρμοσε και εφαρμόζει τα ανακοινοθέντα στη στρατηγική και λαμβάνει μέτρα που δεν προβλεπόταν στρατηγική. Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία για να δείξω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι προτίθεται να κάνει σχετικά με τη διαφορά αμοιβών ανδρών και γυναικών. Το πρώτο που ήθελα να αναφέρω. Το ανέφερε και προλίγου κυρία Μπάουερ. Η εισαγωγή της ημέρας αυτής για την ισότητα των αμοιβών. Αυτή η μέρα σημαίνει μέχρι ποια μέρα πρέπει να δουλέψουν την, ε- τον επόμενο χρόνο οι γυναίκες να συμπληρώσουν την αμοιβή τους για να αντιστοιχεί στην αμοιβή που παίρνουν οι άντρες. Εορτάστηκε, τέλος πάντων, σημειώθηκε για πρώτη φορά το 2011. Θα επαναληφθεί αυτό φέτος, τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα πιο πρόσφατα στοιχεία. Ήταν 5 Μαρτίου το 2011, άρα ελάχιστη η βελτίωση στα στοιχεία Οπότε η μέρα πήγε λίγο πιο μπροστά, 2 Μαρτίου, απαράδεκτη βελτίωση. Σημαντικότατο το εγχείρημα ε, για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη διαφορά των αμοιβών ανδρών και γυναικών. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Δεύτερον, κάτι που δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια μελέτη το 2011 η μελέτη αναλύει ευρύ φάσμα πολιτικών, μέτρων, νομοθετικών και μη νομοθετικών. Αυτά συμπεριλαμβάνουν, κυρίως τα περισσότερα, τις συστάσεις του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου του 2008. Και πολλά από αυτά που στη συζήτηση, μέτρα για την βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τις αμοιβέ, μέτρα όσον αφορά τις κυρώσεις, για διάκριση μη νομοθετικά μέτρα. Παραδείγματο χάρη, πιστοποιητικό για ε, ίσες αμοιβέ, κάτι που αναφέρθηκε, όλα συμπεριλαμβάνονται στι πολιτικές που αναλύσαμε στη μελέτη. Η μελέτη ολοκληρώνεται τώρα, θα ολοκληρωθεί σύντομα, όταν θα είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τι συνέχεια μπορεί να δοθεί σε αυτό το μέτρο. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν και κάτι σημαντικό. Συμπεριλαμβάνεται και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για μελλοντικά ενδεχόμενα μέτρα για να καλυφθεί αυτή η διαφορά των αμοιβών. Είναι στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012. Θεωρείται σαν μια πρωτοβουλία που θα αναλυθεί το 2013. Η διαβούλευση δηλαδή με τους κοινωνικού εταίρους όσον αφορά τη διαφορά των αμοιβών αδών και γυναικών και τα μέτρα που θα ληφθούν για να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Αυτά κάνουμε λοιπόν για την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση έλαβε και ευρύ φάσμα άλλων μέτρων. Ε, εκστρατεία ενημέρωση και πληροφόρηση που αναφέρθηκε στη συζήτηση, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειε. Μόλις ξεκινήσαμε και άλλη πρωτοβουλία, ε, ζητήσαμε υποβολή προσφορών, εκδήλωση ενδιαφέροντων, ενδιαφέροντος, για νέα προσπάθεια ευαισθητοποίηση. Στόχο οι επιχειρήσει. Κυρίω μέσω δραστηριοτήτων κατάρτιση και ανταλλαγή καλών πρακτικών κάποια πράγματα που έγιναν ήδη στην ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών ήταν ότι ετοιμάζαμε εμείς διάφορες ε, διασκέψεις όπου εξετάζαμε συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών. Παράδειγμα. Πολύ θετικό. Η ανάπτυξη λογισμικού που επιτρέπει στους εργοδότες γιατί και οι εργοδότες καμιά φορά δεν γνωρίζουν το βαθμό διαφοράς αμοιβών ανδρών και γυναικών στην εταιρεία τους, δεν το προσέχουν έλεγα ευαισθητοποιούνται οι εργοδότες και μπορούν μέσω του λογισμικού να δουν αυτή τη διαφορά των αμοιβών και να κινηθούν κατάλληλα και μπορούν έτσι ή να μειώσουν τη διαφορά ή να την εξαλείψουν. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό. Αναφέρθηκε επανειλημμένα στη συζήτηση. Τα στατιστικά στοιχεία για τη διαφορά των αμοιβών ανδρών και γυναικών. Είναι πολύ περίπλοκο το φαινόμενο. Συμπλαμβάνεται η διάκριση στο φαινόμενο, αλλά όχι μόνο αυτό γιατί η διάκριση απαγορεύει τους κανόνες τη συνθήκη. Χρειάζονται στατιστικά στοιχεία και η Eurostat θα αλλάξει τον κανονισμό για την κατανομή στοιχείων και θα προσπαθήσει να δώσει καλύτερε πληροφορίε για το πώ αυτή η αλλαγή ε, διαφορά αμοιβών μεταξύ, πώ και γυναικών. Λοιπόν, πέρα από τη ρουτίνα που οφειλεται αυτη η αλλαγη διαφορα αμοιβων να εδω και γυναικων λοιπον περα απο τη σχέση νομοθεσία, Λάβαμε πολλά άλλα μέτρα που καλύπτουν ευρύ φάσμα για να αντιμετωπίσουμε πολυδιάστατη, περιπλοκότατη κατάσταση από διάφορες γωνίες. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια, να εξετάσουμε κάθε δυνατότητα και επικείμενη μελέτη και ανάλυση αυτής και τα συμπεράσματα που θα συναχθούν είναι σημαντικό βήμα. Και κάτι άλλο η ισορροπία των φύλων στη λήψη αποφάσεων στον οικονομικό τομέα. Αναφέρθηκε στη συζήτηση. Γνωρίζετε ότι αποτελεί η προτεραιότητα της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ. Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασιών για φέτος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρθηκε αυτό. Αξίζει να δούμε άμεσα και έμεσα αποτελέσματα του μέτρου αυτού που θα έπρεπε να έχει όσον αφορά τη διαφορά αμοιβών αδών γυναικών, διότι η καλύτερη ισορροπία και ποικιλία των φύλων στους φορείς που αποφασίζουν για τη δομή των επιχειρήσεων του προσωπικού θα είναι ένα σημαντικό βήμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαφορά αμοιβών των γυναικών. Άρα ευρύ φάσμα μέτρων εξετάζουμε. Αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η νομοθεσία είναι μια επιλογή, αλλά όχι μοναδική. Και καμιά φορά ούτε κάνει καλύτερη. Ναι, Κυρία Τσίμερ, να καταλήξετε, γιατί έχουμε ένα τέταρτο καθυστέρηση. Μήπως μπορείτε να τα συνοψίσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ να όλους οι οποίοι έλαβαν το λόγο από τις διαφορετικές πολιτικές ομάδες για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια ευρεία συνένεση σε από, με συμμετοχή όλων των κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να καταλήξουμε σε μια συνεκτική γνωμοθότηση προς το ψήφισμα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Αυτό θα δείξει και την ε, σαφή μας πεποίθηση όλων οι οποίοι έχουν λάβει το λόγο και ζήτησαν να υπάρξει κάποια προσπάθεια για να καλυφθεί αυτό το κενό. Ζητώ από όλους λοιπόν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις και εγώ είμαι στη διάθεσή τους να συνεργαστώ με τις τροπολογίες τους για να δούμε επίσης και τι έχει προκύψει με την ε, οικονομική κρίση και να καταδείξουμε ότι υπάρχουν και περαιτέρω αρνητικά αποτελέσματα από την κρίση. Αυτό που είπε η κυρία Οβίρ από την, Έσλαντ, από την, Ισλανδία, από την Εστονία συγγνώμη, είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλέ από τις χώρες μας όπου βλέπουμε ότι αυξάνεται η διάκριση κατά των γυναικών στον χώρο εργασίας και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Να επιστήσω την προσοχή σας λοιπόν επίσης και στο γεγονός ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλες πτυχές όπως είναι η μη εφαρμογή από την πλευρά της Κομισιόν της αίτηση μας να υπάρξει και ισότης, εργασία, ισότης αμοιβών σε εργασία ίσης αξίας. Γιατί σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει μονάχα η νομοθετική ρύθμιση για ίση εργασία να είναι ίση η αμοιβή και όχι για εργασία ίσης αξίας. Και επομένως σε πολλές χώρες είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια διαμφισβήτηση για το κατά πόσον μια εργασία που είναι ίσης αξίας δεν ε, αμείβεται αντίστοιχα και επομένω υπάρχουν πολλές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και με πρόταση τη Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κλείσει λοιπόν με αυτό το θέμα που ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και επί της βάσης αυτής που αναφέρθηκε θα μας παρουσιάσει η κυρία Τσίμερ. Θα ανοίξουμε καταρχήν την προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου το μεσημέρι και θα τις εξετάσουμε στις 29 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου. Πάμε στο σημείο 20 της ημερησίας ημών διατάξεως και δίνω το λόγο στην κυρία Ίνες Τσιμπέρ για την πρώτη της έκθεση η οποία έχει αναλάβει τη σκητάλη από την κυρία Ιλντε Φίγκερέντου η οποία ήταν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών το 2013 και έχουμε να, έχει να αντιμετωπίσει 90 τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Κυρία Ζουμπέρ έχει το λόγο για να δώσετε ενδείξεις για αυτές τις τροπολογίες λόγω τη καθυστέρηση που έχουμε συσσωρεύσει. Σας παρακαλώ να είστε σχετικά σύντομοι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ σε ως το δυνατό λιγότερο χρόνο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που έχουν καταθέσει τροπολογίες σε σχέση με την πρόταση αυτή, με την γνωμοδότηση αυτή σε σχέση με μια πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <clears throat> σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών το 2013. Είμαι βέβαιη ότι οι προτάσεις αυτές τροπολογίας εμπλουτίζουν το κείμενο της γνωμοδότησης και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις απαραίτητες συμβιβαστικές λύσεις σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση. <clears throat> Έχω κάποια σημειώματα εδώ σε ενδεχόμενες γραμμές συνένεση σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και θα αναφέρω τώρα ότι καταρχήν η ιδέα της ενίσχυσης της Ιταγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ελεύθερης κυκλοφορίας έχει πληγεί από κάποιες μορφές ε, περιορισμών λόγω εθνικότητος, λόγω φύλου, λόγω σεξουαλικής ε, προτίμησης κτλ. Η ελεύθερη αυτή κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρχει πλήρης προστασία των πολιτών στα πλαίσια αυτής της, ε, σε αυτές τις διακρίσεις. Είναι απαραίτητο επίση να υπάρξει και προστασία των εργαζομένων από τρίτε χώρε οι οποίοι διαμένουν στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να απολαμβάνουν και αυτοί και οι οικογένειέ του τα ίδια δικαιώματα με του άλλου εργαζόμενου τη χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να έχουν την ίδια σχέση με τι οικογένειέ του όπω οι εργαζόμενοι τη ε, αντίστοιχη χώρα μέλου όπου εργάζονται. Επίση, Πρέπει να τονίσουμε την αξία της ισότητας, της ε, ελευθερίας και της ασφάλειας που περιλαμβάνονται για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τονίζω επίση το θέμα της κινητικότητας, της εθελοντικής κοινοτικότητας, η οποία μπορεί να αυξήσει και μια καλύτερη σχέση μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω και προγραμμάτων τα οποία προωθούν αυτή την κινητικότητα <clears throat> και επίσης για όλε τι πρωτοβουλίε που φέρνουν σε επαφή πολίτε με διαφορετικέ ηλικίε ή διαφορετικά επίπεδα μόρφωση και επαγγελματικών προσόντων. Είναι επίση σημαντικό να υπάρξει πλήρη παροχή πληροφοριών σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων για την τα δικαιώματά σε σχέση με την προστασία της κοινωνικής ασφάλειας, τα δικαιώματα αμοιβή του, τα, τις συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης. <coughs> και αυτό αφορά και τους εργαζόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτούς που είναι από τρίτες χώρες και διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, είναι απαραίτητο οι πληροφορίες αυτές να δίδονται σε διάφορα υπόβαθρα, ηλεκτρονικά και ε, μη, σε διάφορες γλώσσες και οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να μεταλαμβαδεύονται μέσω των κοινωνικών εταίρων. και το πρόγραμμα EURES <coughs> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια καλύτερη παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. Τονίζω επίσης την ιδέα ότι τα κοινωνικά, τα συνδικαλιστικά και τα εργασιακά δικαιώματα θα πρέπει να, να τύχουν προάσπισης, να μην παρακάμπτονται και να υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων και να μην <clears throat> ευνοούνται ε, καταστάσεις που οδηγούν στην λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων και στην πορνεία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλιστεί το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, παιδείας και απολαβής κοινωνικών παροχών. Επίσης, έχω τονίσει την ανάγκη να ξεπεραστούν τα διοικητικά και νομικά εμπόδια που πλήττουν τους πολίτες που θέλουν να ζήσουν σε άλλο κράτος μέρος. Και επίσης αναφέρω τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με εθνικότητα, κοινωνικό ή <clears throat> οικογενειακό πλαίσιο κτλ. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι αυτοί οι περιορισμοί οδηγούν πολλές φορές στην παράνομη εργασία, στην αύξηση της παράνομης εργασίας με αντικό αποτέλεσμα και για τους εργαζομένους και για τις κοινωνίες όπου διαμένουν. Αυτά λοιπόν είναι διάφορα σημεία που διατρέχουν την ε, <clears throat> πρόθεσή μου για το έγγραφο εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για τη βοήθεια που μου έχουν δώσει κατά την εκπόνηση αυτού του εγγράφου. Ευχαριστώ. Σας κατευχαριστώ. Κυρία Σιπέλ και μετά Μαρκή. Ε, ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν την ε, αρχική εισηγητρία, την κυρία Φιγκέι Φιγκέιρέντο, η οποία έχει αφήσει μια πολύ καλή γνωμοδότηση και να ευχαριστήσω και την κυρία Ζούπερ με την οποία μπορέσαμε να είχαμε ήδη μια πολύ επωφελή συνεργασία την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορώ να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε η κυρία Ζούμπερ ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες οι οποίες έχουν την ίδια κατεύθυνση ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδος θέλουν να τονίσουν την ανάγκη της καταπολέμησης των ε, ε, <clears throat> διακρίσεων, τη ίση μεταχείρισης, αντιμετώπιση αντιμετώπισης μειονεκτικών ομάδων, τη καλύτερη κινητικότητα. Όλα αυτά είναι στοιχεία λοιπόν τα οποία μπορούν να καλυφθούν από κοινέ συμβιβαστικέ τροπολογίε. Θέλω να αναφέρω όμω και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο αναφέραμε και σε προηγούμενε οδηγίε, <clears throat> το γεγονό ότι υπάρχει μια σταδιακή αποδόμηση των δικαιωμάτων και τα κεκτημένα των πολιτών, τα δικαιώματα των πολιτών βρίσκονται ε, <clears throat> σε κατάσταση μείωσης και διάβρωσης και πολλές φορές και οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν αυτά τα δικαιώματα και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για να διατηρήσουμε αυτά τα κεκτημένα των πολιτών και να τα κάνουμε γνωστά σε αυτούς. Υπάρχουν κάποιες ορισμένες ε, τροπολογίες που είναι κάπως προβληματικές. Αυτά τα οποία <coughs> αφορούν τα μέσα ενημέρωσης και επίσης σε σχέση με μια έκθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα είναι ίσως δύσκολο να αναφερθούμε σε αυτά τα θέματα όταν υπάρχει ήδη μια ζωντανή συζήτηση για τα, την ελευθερία των μέσων επιχειρήσεων. Κάτι άλλο που μας αφορά είναι η λεγόμενη διαρροή εγκεφάλων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η κατάλληλη κατάρτιση των πολιτών στις χώρες μας. Δεν θέλουμε η κατάρτιση αυτή να τους οδηγήσει εκτός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, θα θέλαμε να ευνοήσουμε την ε, εισρωή εγκεφάλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες χώρες, η οποία οδηγεί σε λιγότερα προβλήματα. Επίσης, είναι χρήσιμο να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών για την ε, ύπαρξη θέσεων απασχόλησης και έτσι η διαδικτυακή θύρα Εύρες μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε αυτό και να προσθεθούν και άλλες διαδικτυακές θύρες. Η τροπολογία 89 της κυρίας Φιγκερέντο επίση τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει και δυνατότητα μεγαλύτερης δημοσιότητας σε συνδιασκέψεις σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά επίσης να υπάρξει και προσπάθεια να καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία και η πορνεία στους μετανάστες από τρίτες χώρες. Λοιπόν, εάν αναφερόμαστε σαν Επιτροπή Απασχόλησης στα θέματα αυτά, θα πρέπει να ζητήσουμε η σύνολη προβληματική της μαύρης εργασίας να αντιμετωπιστεί ε, συνολικά και από τα κράτη-μέλη και όχι απλώς σε επίπεδο πληροφόρησης των πολιτών και των εργαζομένων. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε περαιτέρω επιτυχή και θετική ε, συνεργασία με την κυρία Ζούμπερ, γιατί είναι απαραίτητο για το έτος αυτό να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν τα κεκτημένα των εργαζομένων. Μαρκή Μπεκέρ και θα τελειώσουμε με άλλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φιγκερέιντο για της για την εξαιρετική της έκθεση και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά και με την διάδοχό της. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους μετανάστες και τις οικογένειές τους, πρέπει να καταλάβουμε ότι η κινητικότητα των εργαζομένων δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μειονέκτημα, όπως είπε το πρωί και η εκπρόσωπο της Δανικής Προεδρίας. Δεν κινούνται απλώς για να κινηθούν, αλλά και για να σπουδάσουν, για να εργαστούν κλπ. Και αυτό το δικαίωμα το έχουν από την ευρωπαϊκή τους ηθαγένεια. Υπάρχουν μια-δυο τροπολογίες πολύ χρήσιμες ότι όλοι αυτοί δεν πρέπει απλώς να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα να τα ασκήσουν. Υπάρχουν και μερικές άλλες για την άνηση μεταχείριση, με βάση την πρωτοβουλία των πολιτών και τα ατομικά δικαιώματα. Τα, αυτά αναφέρονται βέβαια στη χάρτα των θεμελιωδών. Επίσης υπάρχουν μία-δύο όπου λέμε ότι δεν υπάρχει μόνο δικαίωμα συμμετοχή στην πολιτική ζωή αλλά και διαμόρφωσης και έκφρασης απόψεων και προσφυγής στον διαμεσολαβητή. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Λίγες είναι οι τροπολογίες που ξεπερνούν κατά πολύ τις ιδέες της Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι η έκθεση της κυρίας Φιγκερέντο είναι πολύτιμη γιατί καταλήγει στο ότι σε συνένεση μεταξύ μας για τα περισσότερα σημεία της διότι η συμπερίληψη της πρωτοβουλίας των πολιτών είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και με ενδιαφέρει πολύ, πολύ η πρόταση αυτή. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε ένα λάθος που ήδη έγινε στο παρελθόν Ξέρετε ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Δεν έχουμε. Και ένα από τα προβλήματα είναι ακριβώς η έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών για τα δικαιώματά τους. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος επικοινωνεί με ποια μέσα και με τι αποτελεσματικότητα. Αυτά έχουν μείνει αναπάντητα νομίζω και πρέπει να τα απαντήσουμε. Με χαρά διαπιστώνω ότι μερικές τροπολογίες το θέτουν αυτό το πρόβλημα και δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε την ουσία αν οι πολίτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Πολλές φορές δεν ξέρουν καν ότι έχουν ευρωπαϊκή ηθαγένεια, ότι είναι πολίτες της Ευρώπης ή τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνουν όπως εμείς. Αυτό είναι δικό μας καθήκον της Επιτροπής μας να τους ευαισθητοποιήσουμε για αυτό το θέμα. Η ευθύνη των χωρών μελών επίσης είναι αδιαμφισβήτητη και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης επίσης πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο. Υπάρχει και μια παρεξήγηση στο σημείο 4 όπου νομίζω ότι υπάρχει ένα λαθάκι γιατί δεν επιτάσσουμε τίποτα προς τα μέσα. Λέμε απλώς ότι πρέπει να γνωστοποιούν για την ύπαρξη των κυριατέρων θεμάτων και να τα μεταφέρουμε στα μέσα, να γνωστοποιούμε. Μάλιστα, η συγγήτρια. Ευχαριστώ τους πάντες και τις πάσες. θα κάνω συμβιβαστικές προτάσεις για τις τροπολογίες με βάση τη συζήτηση που έγινε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάει και αυτό λοιπόν. Και τώρα φτάνουμε. Τώρα ξέρω ότι η συγγήτριά μας θα μας καταθέσει τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Τις εξετάσουμε 29 Φεβρουαρίου του Αγίου Κασιανού και θα τις ψηφίσουμε την 1η Μαρτίου. Η ΔΕ Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών θα ψηφίσει στις 12 Απριλίου. Ερχόμαστε τώρα στο πρώτο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης λόγω των τροποποιήσεων που δεχτήκαμε το πρωί. Το 21 η κυρία Μορέν για την εξέταση 233 τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στην έκθεσή τη για τι ελάχιστε προδιαγραφέ ασφάλεια και υγεία όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνου προερχόμενου από φυσικού παράγοντε παρένθεση ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ορίστε κυρία εισηγητρία, έχετε τον λόγο. Πρέπει απλώς να σας πω ότι υπάρχει μια δυσκολιούλα γιατί η συντηρητική, για τους συντηρητικούς η κυρία Τζούλια Γκίρλινγκ ήταν η εισηγήτρια, ήταν ε, σκιώδης μάλλον δεν είναι όμως πλέον μέλος της Επιτροπής μας. Φυσικά μπορεί να συμμετάσχει όπως όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά επισήμως, επισήμως δεν μπορεί να είναι σκιώδης. Πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον της ομάδας της. Ορίστε κυρία εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι υπάρχουν 233 τροπολογίες πολλές από τις οποίες, γιατί 91 είναι από τους πράσινους και οι υπόλοιπες κατανέμονται λίγο πολύ σε όλες τις ομάδες, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέταξαν από τους σοσιαλιστές τη Σιλβάνα Ράπτη, την Καρή Μαντελή από τους Πράσινους, από τους φιλελεύθερους την Λίζ Λίν που τη χαιρετίζω εδώ και εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία της κυρίας Γκυλίνγκ που ήταν μέχρι πριν από λίγο σκιώδης συγγήτρια για τους συντηρητικούς και τον κύριο Τούσα από την ΚΟΕ. Η συνεργασία μας ήταν έγινε μέσω πολλών συνεντήσεων και κάθε ομάδα μετά κατέθεσε τις τροπολογίες της όπως φρονούσε. Πάντως τα γενικά πλαίσια μας υποχρεώνουν να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμασταν μέχρι τώρα με την οδηγία αυτή από το 2004 που δεν μπόρεσε ακόμη να εφαρμοστεί. Η εφαρμογή της αναβλήθηκε για τις 30 Απριλίου φέτος, πράγμα το οποίο μας υποχρεώνει να καταλήξουμε σε ένα νέο κείμενο, μια νέα οδηγία που να είναι εφαρμόσιμη αυτή τη φορά που να είναι βιώσιμη και άρα και που να λαμβάνει υπόψη της τις απαραίτητες εξαιρέσεις διότι δεν μπορούσε να εφαρμοστεί ιδιαίτερα στον ιατρικό τομέα για τις, για τις μαγνητικές αντιχήσεις γιατί εκεί για ορισμένες αρρώστιες χρειάζονται εξαιρέσεις ιδιαίτερα όσον αφορά καρκίνους και άλλες εκφυλιστικές ασθένειες νευρολογικού κυρίως χαρακτήρα. Έχει γίνει λοιπόν μία αναπροσαρμογή της οδηγίας του 2004 που ήταν ανεφάρμοστη ως είχε, ώστε να καταλήξουμε σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση που να προστατεύει την υγεία των εργαζομένων που υφίστανται ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά επίσης να διατηρεί την ύπαρξή τους για ιατρικούς λόγους, για ιατρικούς ελέγχους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί να εξισορροπήσουμε το κείμενο. Και θέλουμε για τους εργαζόμενους να, γίνει μια, να γίνεται μια τακτική επανεξέταση της οδηγίας για να βλέπουμε τι από όσα λέμε δεν έχει απολύτω επιστημονικά ελεγχθεί και να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις της επιστήμης αν χρειαστεί. Ορισμένες τροπολογίες έχουν κατατεθεί για αυτόν τον σκοπό που ζητάει αυτή την τακτική ανα... επανεξέταση κάθε πέντε χρόνια. Δεύτερον σημαντικό θέμα. Οι τροπολογίες πολλές από τις τροπολογίες μιλούν για την ανάγκη να υπάρχουν είπα αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για ιατρικούς σκοπούς ε, Νομίζω ότι θα βρεθεί μια συνένεση, κανείς από εμά δεν θα ήθελε να υποστεί μια νόσο που να χρειάζεται μαγνητική αντίχηση αλλά να μην μπορεί να την κάνει ο γιατρός, να με απαγορεύεται δηλαδή. Κανείς δεν θα ήθελε να στερηθεί της εξέτασης αυτής. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τρίτον, θέμα επί του οποίου υπήρξαν διαμάχες και διαφωνίες μεταξύ των ομάδων οι επιπτώσεις, ορισμένοι λένε οι πιθανές επιπτώσεις, αλλά γιατί καμία δεν έχει αποδειχτεί, οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Τέταρτον, σημαντικό θέμα που θίγουν οι τροπολογίες, η αναγκαιότητα να υπάρχει μία πληροφόρηση και επιμόρφωση όσων εργάζονται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και κάτι που νομίζω προκύπτει από το πρώτο, η ανάγκη να γενικευτούν οι βέλτιστες πρακτικές. Και οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να συσταθούν για την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των πεδίων αυτών. Τέλος, μερικοί προτείνουν όρια έκθεσης, ημερήσια όρια έκθεσης, αλλά καταλαβαίνετε ότι γενικά πρόκειται για πολύ περιορισμένες εκθέσεις σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έλαβα και ένα γράμμα της κυρίας Καρίμας Δελή που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα που λίγο πολύ ή μάλλον ούτε λίγο ούτε πολύ ε, από τι φόρο τιμής στην Επιτροπή μας και στην ομάδα εργασίας μας μάλλον και που συμφωνεί ότι πρέπει να συνδυαστεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων με, με την ιατρική περίθαλψη και κάνει προτάσεις τέτοιου είδους. Μόνο επ' αυτού θέλει να επιμείνει σήμερα στην επιστολή της. Τις υπόλοιπες τροπολογίες που προτείνει για τις υπόλοιπες δεν επιμένει, δεν τις αναφέρει καν σε αυτή την επιστολή. Τέλος, πάλι, θα ήθελα να σας πω ότι με τις διαβουλεύσεις που έκανα είδα ότι όλοι υφιστάμεθα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όλοι εκτιθέμεθα, αλλά ορισμένοι, ορισμένα από αυτά είναι πολύ ισχυρά και δεν τα προσέχουμε όπως κύριοι, τα ηλεκτρικά ξηράφια, οι ηλεκτρικές ξηριστικές μηχανές ή τα σεσουάρ κυρίες μου. Ας μην πανικοβαλόμεθα όμως. Ξέρουμε ότι υπάρχει και το θέμα της υγείας των εργαζομένων, ότι υπάρχουν πολλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία αλλά και ότι δεν πρέπει να υπάρξει πανικός επ' αυτών. Γιατί μας ωφελούν και όλα στην υγεία. Ευχαριστώ. Ε, Λίν. Η κυρία Λίν, σας χαιρετίζω, χαίρομαι που είστε εδώ. Νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες φορές που θα σας δώσω το λόγο. Και η κυρία Ράπτη μετά. Πρώτα κυρία Λίν. Ευχαριστώ. Ναι, αποχωρώ το τέλος επόμενης εβδομάδες και θα κάνω και ένα πάρτι 1η Φεβρουαρίου για την αναχωρησή μου, οπότε μπορείτε σε 6.30 να έρθετε κάποιοι από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίζαμπεθ, για τη δουλειά που έκανες. Ε, την εκτιμώ. Όλοι μας άλλωστε την εκτιμούμε. Πολύ καλή έκθεση που συνέγραψες και ελπίζω να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα οι τροπολογίε που υπευλήθησαν, που υπεύαλα Από το 2004 επεξεργάστηκα το θέμα και χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει διαφορετικό συνέστημα επικρατεί στην Επιτροπή ενώ το 2004 ήμουνα ίσως η μόνη που ήθελε να απομακρυνθεί κάπως από την εντολή της ε, οδηγίας και να προχωρήσει από πέρα. Φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που το θέλει όλη η Επιτροπή και χαίρομαι πολύ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, πρέπει να προσέξουμε αυτά τα εγκεφαλογραφήματα, αυτές τις εξετάσεις που είναι εκτός των ορίων. Θέλαμε να είναι εκτός της οδηγίας αυτές οι εξετάσεις με μαγνητικές ε, τομογραφίες κλπ. Από τη στιγμή θα το κάνουμε αυτό, ε, θα, επί... θα είναι εκτός των οριακών τιμών αυτές οι εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, ούτω ώστε οι σαρωτές υψηλής τεχνολογίας να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αν δεν χρησιμοποιούνται ε, στο μέλλον θα δούμε πολλούς θανάτους παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρη από αυτό βραχυπρόθεσμα, μακρυπρόθεσμα αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε τα βραχυπρόθεσμα. Δεν ξέρουμε τα μακροπρόθεσμα. Καταλαβαίνω στις τροπολογίες που ευλήθησαν, που έλεγαν στο μέλλον πρέπει να συμπεριλάβουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι αν γίνει αναθεώρηση των νέων επιστημονικών στοιχείων, που ίσως διαφανούν για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αυτό είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε προσεκτικότατα, διότι αν ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμε συνέπειε και υπάρχει επιστημονική βάση για αυτό το πόρισμα, θα πρέπει να επανεξετάσουμε την κατάσταση. Δεν νομίζω όμω ότι αυτομάτω θα πρέπει να εξετάζονται αν τα επιστημονικά στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι οι μακροπρόθεσμε συνέπειε αποτελούν πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και να μην δημιουργηθεί, συσταθεί νέα οδηγία για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτομάτω, εκτό αν είναι απόλυτα αναγκαίο κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να έχουμε παράταση του μορατόριου για την ώρα. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε. Συγκεκριμένε τροπολογίε αναφέρω που υπέβαλα. 69. Αφορά τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα. Σε πολλές άλλες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίναμε και που έγιναν νομοθεσία, ξέρουμε ότι ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι ασφαλής. Οι σαρωτές πρέπει να είναι ασφαλής και πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις για τους κατασκευαστές των μηχανημάτων. Εξού και η τροπολογία μου. Τροπολογία 79. Την είχα υποβάλει όταν το συζητήσαν το θέμα. Δεν είναι μόνο οι χειριστέ των μηχανημάτων, είναι οι ερευνητέ, οι καθαριστέ, το προσωπικό, οι συντηρητέ. Πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τροπολογία 146. για το ωκεάνιο θα έπρεπε να υπάρχει είτε ξεπερνούνται οι ε, οριακές τιμές είτε όχι. Φαίνεται γελίο. Στον τομέα αυτό ενδεχομένω, εάν δεν χρειάζεται ε, να ξεπεραστούν τα όρια, δεν κάνουμε κάτι. Αν ξεπερνούνται τα όρια θα πούμε ότι οι οριακές τιμές πρέπει να τηρούνται. 146 τροπολογία. Εκπαίδευση των εργαζομένων. Σημαντικότατο. Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Εκπαίδευση επαρκής για εκείνους που ασχολούνται. Γι' αυτό επέβαλα πολλές τροπολογίες για την κατάρτιση. 151. Συμφωνείτε, ξέρω με πολλά από αυτά που θέτω. Αλλά για την υπόλοιπη επιτροπή λέω για ποιους λόγους υποβάζει τροπολογίες. 151 λοιπόν. Πήγα στο αρχικό κείμενο πρέπει να δηλώνουν ότι είναι ε, έγκυοι ή ότι έχουν κάποιες ε, ιατρικές συσκευέ πάνω τους. Καμιά φορά ο εργοδότης δεν επιτρέπεται σε κάποιες περιπτώσεις να ρωτήσει αν είναι έγκυος υπάλληλο ή αν έχει κάποιο ιατρικό, ιατρική συσκευή ε, που χρησιμοποιεί. Λοιπόν, εάν έχει δηλώσει η εργαζόμενη ότι είναι έγκυος ή ότι χρησιμοποιεί κάποια ιατρική συσκευή που είναι πάνω της, πάνω του, πρέπει να δηλώνεται. 160. Έλεγχος της υγείας. Κάλυψε εθνικό δίκαιο και πρακτικές. Διότι ο έλεγχος αφορά την υγεία διενεργείται από τους εργοδότες, καμιά φορά σε κάποια κράτη-μέλη, καμιά φορά πληρώνουν οι κυβερνήσεις σε άλλες χώρες, άρα το ρυθμίζει η εθνική νομοθεσία. Έλεγχος υγειονομικός υγείας, πολύ σημαντικό να καλύπτουν όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι επιτέλους θα περάσει η έκθεση έκθεση η οποία θα προστατεύει τους εργαζομένους και δεν θα είναι δύσκολο να εφαρμόζεται τους εργοδότες από την άλλη. Το σημαντικότερο. Οι σαρωτές, οι μαγνητικοί, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των οριακών τιμών. Και αυτή πρέπει να είναι η βάση, το όριο. Όπως είπα στην αρχή και όπως έλεγε το 2004, εάν δεν το κάνουμε αυτό, και ευτυχώς που άκουσε τη λογική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάλει το μορατόριο Εάν δεν είχε το μορατόριο, οι σαρωτέ, οι μαγνητικοί τομογράφοι δεν θα χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Α ελπίσουμε ότι θα έχουμε τελικά στα χέρια μα μια λογική οδηγία. Καλή τύχη λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή ακόμα και μετά την αποχώρησή μου, το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, καλή τύχη με το όλο θέμα, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ράπτη και μετά και ο Σκλάρκη. Η κυρία Ράπτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εισηγήτρια, την ε, κυρία Σαρτιέ, για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Να την ευχαριστήσω επίσης για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ε, να προσθέσω όμως τον προβληματισμό μου για το παράδειγμα του Σεσουάρ για τα μαλλιά που ανέφερε. Ε, σκέπτομαι ότι στην αίθουσα όλες οι γυναίκες ε, θα σκεφτήκαμε πόσο συχνά στεγνώνουμε τα μαλλιά μας με το σεσουάρ και τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να ανοίξουμε μία ε, ε, ένα άλλο κεφάλαιο για τις συνθήκες εργασίας των κομωτών και των κομωτριών, για το πόσο συχνά πρέπει <laughs> να πηγαίνουμε κομωτήριο και βεβαίως βλέπω τον καλό μου συνάδελφο τον Όλε Κρίστενσεν που σκέφτεται και τα ηλεκτρικά, πώς τα λένε, το ηλεκτρικό ξύρισμα. Κυρία Σαρτιέ, βάλατε ένα καινούριο θέμα στην ατζέντα. Μια καινούρια οδηγία νομίζω χρειάζεται. Λοιπόν, ε, οι τροπολογίες που έχουμε καταθέσει ε, στην έκθεση αυτή ε, μαζί με τον καλό μου συνάδελφο και πάρα πάρα πάρα πολύ έμπειρο σε αυτό το θέμα τον Στίβε Χιούς, είναι βετεράνος στο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και είναι τιμή μου και χαρά μου που συνέβαλε καθοριστικά στη δουλειά που κάναμε. Οι τροπολογίες αυτές λοιπόν είχαν τρεις στόχους για μας. Ο πρώτος στόχος είναι να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και οι ερευνητές με περισσότερα μέτρα πρόληψης όπου αυτό χρειάζεται. Ο δεύτερος στόχος είναι οι ασθενείς, ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ομάδες ασθενών, όπως παιδιά και άνθρωποι με νοητική στέρηση, να μπορούν να υποβάλλονται σε εξετάσεις που μπορούν να χαρτογραφηθούν μόνο με την τεχνολογία των μαγνητικών τομογράφων, μόνο με το MRI. Και τρίτον, να επαγρυπνούμε συνεχώς για νέα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία ενδεχομένως θα απαιτούν αναθεώρηση της οδηγίας που συζητούμε τώρα. Προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένα τέσσερα πράγματα, τα λέω πάρα πολύ ε, συνοπτικά. Ε, πρώτο, προτείνουμε να διαγραφεί η αναφορά που γίνεται στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δεν θα εξηγήσω το γιατί, διότι οι προλαλήσασες το ανέφεραν. Ε, θα προσθέσω μόνο ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αδιάσυστες επιστημονικές έρευνες που να μας πιστοποιούν ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία βάση προστασίας που θα παρέχεται από την οδηγία πλαίσιο του 1989. Ε, δεύτερον, ζητούμε να επαναξιολογηθεί η παρούσα οδηγία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας οποιαδήποτε νέα στοιχεία για την προστασία των εργαζομένων. Τρίτον, εκεί που επιτρέπονται εξαιρέσεις. Παράδειγμα, το νοσηλευτικό προσωπικό που πρέπει να βρίσκεται κοντά στους ασθενείς για την πραγματοποίηση των εξετάσεων ή το στρατιωτικό προσωπικό, για λόγους εξαιρέσεων στο στρατό, να είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα προστασίας και παράλληλα να δίνουν σαφείς οδηγίες για το χειρισμό των μηχανημάτων. Τέταρτον, δεν θέλουμε να επιτρέπεται η έκθεση πάνω από τις οριακές τιμές. Σε όλα αυτά τα ζητήματα ασφαλώς θέλω να ακούσω τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κλείνοντας, ε, κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο χρονοδιάγραμμα. Είναι κάτι που και η Ελιζαμπέτ το είπε με τον τρόπο της. Ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ξέρουμε και οι παλιότεροι το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι το θέμα δεν είναι μόνο να συντάσουμε ψηφίσματα, να τα ψηφίζουμε και να νιώθουμε υπερηφάνεια που τα ψηφίσαμε. Το θέμα είναι αυτά που αποφασίζουμε να γίνονται πράξεις ώστε πραγματικά να έχουν ωφέλεια οι Ευρωπαίοι πολίτες. Έτσι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Περιμένουμε τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράταση της υπάρχουσας οδηγίας για δύο ακόμα χρόνια. Τότε όμως αναρωτιέμαι γιατί αγωνιζόμαστε να τελειώσουμε εδώ τις διαπραγματεύσεις μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ε, προτείνω λοιπόν, ακολουθώντας την Ελιζαμπέτ, να συμφωνήσουμε ενδεχομένως στον ένα χρόνο. Δηλαδή τόσο όσο θα χρειαστούμε, τόσο υπολογίζουμε, ένα χρόνο θα χρειαστούμε για να, να... να ολοκληρώσουμε με όλα τα θεσμικά όργανα τις διαπραγματεύσεις μας. Γιατί διαφορετικά ε, οι εργαζόμενοι θα είναι στο κενό. Και νομίζω ότι αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους όπως λαμβάνουμε ε, πρόνοια να προστατεύονται και οι ασθενείς. Σας ευχαριστώ και βάζω τελεία. Merci. Euh, ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάρκ και μετά ο κύριος Έλμερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε υπενθυμίσω αυτά που είπαν διδικοί από τον Μπάρς και τον Σεντόμα από το Λονδίνο, που μίλησαν πριν από 6 χρόνια σε αυτή την επιτροπή και δεν ήταν ευχαριστημένοι τα όρια για τους αρωτές MRI, είχαν πολύ χαμηλά, ούτω ώστε να αποκλείονται αυτοί οι αρωτές, οι μαγνητικοί τομογράφοι. Και, ρω... και σήμερα, αν ήταν παρόντες θα ήταν ικανοποιημένοι, ρώτησα. Και μου είπαν ότι θα ήταν. Οπότε στέλνω αντίγραφο του 40... των 40 σελίδων του χειριδίου τότε στο βασιλικό ε, ε, σώμα των χειρούργων και της αδειογραφίας για να ρωτήσω κατά πόσο είναι όλα καλά. Και ένας από τους πυρογνώμονες, ο Dr. Κίφελ του King's College, ήταν στις Βρυξέλλες σήμερα και μου έδωσε μισή ώρα μου έθεσε. Και τον ρώτησα το ίδιο πράγμα. Και είπε ναι, θα ήταν ικανοποιημένο. Ε, οι οριακέ τιμέ τώρα έχουν ξανατοποθετήσει σε απόδεκτο επίπεδο για του τομογράφου, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που αναμειγνύονται. Ιδιαίτερα ήθελε η Επιτροπή να παραδεχτεί και να υιοθετήσει τα παρατήματα 3 και 4 που θα πρέπει απλώς να περάσουν. Διότι βλέπετε συμπεριλαμβάνουν παρεκκλήσεις που υπευλήθησαν πιστεύω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιτρέπουν το θεατρικό προσωπικό σε κάποιες περιστάσεις να παραμείνει με τον ασθενή κατά τη διάρκεια της χρήσης του σαρωτού, όταν γίνεται σάρωση. Τότε οι ασθενείς είναι αυτοί που έχουν κάποιο πρόβλημα ε, νέα παιδιά που είναι νευρικά, έχουν άγχο και λοιπά και το καταλαβαίνω. Έπρεπε πριν από ένα μήνα να κάνω μια σάρωση και οι 20 λεπτά θα πρέπει να παραμείνει ακίνητο ενώ ακού θόρυβο από τον τομογράφο, κάνει παράξενου θορύβου γύρω ο τομογράφο και τα νέα παιδιά θα έπρεπε να δέχονται την ανακούφιση και τον καθησυχασμό από το ιατρικό προσωπικό, όπω και κάποια άνθρωποι που έχουν κάποια πνευματικά προβλήματα, γενετικά προβλήματα, φυσικά προβλήματα και κάποιοι ασθενεί ε, δέχονται περαιτέρω θεραπεία κατά τη διάρκεια της άρρωσης ενώ γίνεται η άρρωση. Άρα είναι ζωτική σημασία, κυρία Πρόεδρε, αυτό. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις το ιατρικό προσωπικό να είναι ε, στην ίδια αίθουσα όπου είναι και η συσκευή άρρωση τη στιγμή που σαρώνεται ο ασθενή Και παρακαλώ η Επιτροπή να υποστηρίξει συνεπώ τα παρατήματα και τέσσερα πλήρω και απολύτω. Και αν αυτό συμβεί, όπω το βλέπω, αυτή η έκθεση θα ε, είναι μια χαρά. Θα είναι αυτό που πρέπει ο κύριος Έλμερ και η κυρία Εγκέρινγκ μετά. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επιτρέπετε να ρωτήσω κατά πόσο συνάδελφός μου κυρία Γκέρλινγκ μπορεί να μιλήσει πρώτα διότι ήταν σκιώδης για την έκθεση αυτή εκ μέρους της ε, ομάδας μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρασία για τη συνεργασία της. Ε, ελπίζω ότι θα συνεχιστεί το πνεύμα συνεργασίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα ε, και έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να πετύχουμε το στόχο μας, να τα κάνουμε όλα σωστά. Ελπίζω ότι θα τα κάνουμε σωστά. Ε, εγώ ανησυχώ μήπως καθυστερήσουμε. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Ε, περιπλοκότατο είναι το θέμα αυτό. Ήταν πρόκληση για όλους. Είναι μια πρόκληση. Ε, και αυτό είναι που το κάνει τόσο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε. Ε, υπάρχουν δύο απλές ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι για του εργαζομένου και ποιο είναι ο πιο ενδεδειγμένο τρόπο για να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύονται οι εργαζόμενοι από του κινδύνου. Ε, υπέβαλα διάφορες τροπολογίες που ελπίζω ότι θα γίνουν θετικά δεκτέ. Η πρόταση αντικατοπτρίζει τη δουλειά που έκανε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για τι συνέπειε των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, συνέπειε που έχουν στο ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιεί εκτεταμένα στοιχεία που έχει παράγει έρευνα και αποφεύγονται τα αρχικά θέματα, περιέχει η αρχική οδηγία όμως. Και όταν διαβάζετε κάποιες τροπολογίες βλέπετε ότι έχασαν το στόχο. Λυσμονήθηκαν τα επιστημονικά στοιχεία και η προσέγγιση που ακολουθήθηκε βάσει των επιστημονικών στοιχείων βασίζονται σε κάποιε εικασίε, υποθέσει, προλήψει θα έλεγα, αλλά είναι λίγο άδικο να λέω προλήψει. Αυτή η οδηγία πραγματικά θα πρέπει να εδράζεται επί συγκεκριμένων στέρεων επιστημονικών στοιχείων και έρευνα. Άρα θα πρέπει να είναι ηλίου φαϊνότερο ότι εξετάζονται τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και μόνο. Ε, πολλές από τις τροπολογίες ε, που είδαμε ζητούν αναθεωρήσεις. Ε, στο πνεύμα συνεργασίας θα μπορούσα να σκεφτώ αναθεωρήσεις επανεξέταση και αξιολόγηση νέων στοιχείων σε πέντε χρόνια. Πρέπει να συμφωνήσω με την κυρία Λίν που είπε ότι θα ήταν εσφαλμένο απόλυτα λάθος τώρα να ζητήσουμε νέες ρυθμίσεις, νέα οδηγία σε πέντε χρόνια. Προϋποθέτει αυτό σωρία ε, αποδείξεων και στοιχείων που ίσως να μην εμφανιστούν, να μην υφίστανται τελικά. Και παίζουμε την ιδέα ότι κάτι υπάρχει που δεν ξέρουμε και ακόμα δεν το έχουμε αναγνωρίσει, δεν το έχουμε δει ακόμα. Και αυτή είναι η εσφαλμένη προσέγγιση όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να είμαι πραγματιστέ όταν συντάσσουμε τη θέση μα τι επόμενε εβδομάδε. Θέλουμε τελικά να έχουμε μια οδηγία που θα είναι αποτελεσματική και θα υπάρχει συμμόρφωση και εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, λέγω. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζω πλήρω την προτινόμενη προς, ε, παρέκκληση για τομέα των μαγνητικών τομογράφων. Κύριε Κλάρ και εγώ πέρασα αυτή τη άρρωση. Δεν είναι πολύ ευχαρίστω, αλλά χαίρομαι που υπάρχει αυτή η τεχνολογία διότι μπορεί να πετυχαίνει κάποια υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και το πεδίο της παρέκκλησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις ιατρικές διαδικασίες διαδικασίε υποστήριξη, ε, υποστήριξη, σύντηρηση, ανάπτυξη, προστασία του προσωπικού. Για την ομάδα μου αυτό είναι κρισίμου σημασία. Είμαι στεναρά κατά εσδήποτε τροπολογίε που προσπαθεί να αφαιρέσει την εξαίρεση και υπάρχουν πάρα πολλέ τροπολογίε που θέλουν αυτό. Και είμαι κατά εσδήποτε τροπολογίε που θέλει να αφαιρέσει εξαίρεση για άλλε ειδικευμένε δραστηριότητε όπω ένοπλε δυνάμει. Εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τεράστια πρόκληση μπροστά μα. Λυπούμε που σε αυτή τη φάση εγώ βγάζω την ουρά μου από μέσα. Ε, η κυρία Μάκενταρ που είναι εδώ η συνάδελφός μου θα αναλάβει τη σκητάλη ε, η, γραμματεία θα κρίνει πρέπει να αλλάξουμε τα ονόματα κλπ αυτά είναι μικρολεπτομέρειες αλλά περιμένει πως και πως να συνεργαστεί με τους υπολείπους σε αυτό το θέμα ευχαριστώ ο κύριος Έλμερ έχει τώρα το λόγο κοιτάξτε σας έδωσα το λόγο πρώτα είχατε σηκώσει το δάχτυλο πριν ε? δεν ήθελα να παρέμβω τέλο πάντων με τι υποθέσει σα, το θέμα σα. Έλμερ Τόμας Μάν, τελευταίος. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Έλμερ είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Κυρία, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι πράγματι πιστεύω ότι έχω μείνει στα κρύα του λουτρού, ότι έχω μείνει απ' έξω και νιώθω ότι έχω υποστεί αντικές διακρίσει γιατί ποτέ δεν πέρασα σαρωτή μαγνητική απεικόνηση δια συντονισμού. Νομίζω ότι όλες οι παρατηρήσεις έχουν γίνει από τους συναδέλφους και έχουν τονιστεί και πολλές φορές. Αλλά ε, θα ήθελα να ρισκάρω να υπονομεύσω την ε, φήμη της κυρίας Λίν λέγοντας ότι συμφωνώ 100% με όλα αυτά που λέει. Συμφωνώ λοιπόν για την εξαίρεση των, ε, μαγνητικών, των σαρατών μαγνητικού συντονισμού και έχω λάβει πάρα πολλές επιστολές από τον ιατρικό χώρο που μου ζητούν να υπάρξει αυτή η εξαίρεση και επίσης είναι η ανάγκη να λάβουμε υπόψη και τις βραχυχρόνιες και όχι μόνο τις μακροχρόνιες εκθέσεις σε μαγνητικά πεδία. Ένα σχόλιο ακόμα. Μου φαίνεται ότι προτείνουμε να κάνουμε αυτή την εξαίρεση για τους σαρωτές μαγνητικού συντονισμού γιατί εμείς ξέρουμε ότι οι μη οι δήμονες μπορούν να καταλάβουν τη σημασία αυτή τη τεχνική. Έχουμε καταλάβει ότι οι κίνδυνοι του να μην υποβάλτηκαν σε τέτοιου είδου τομογραφία είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο της τομογραφία. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες εφαρμογές είτε στην ε, ιατρική είτε σε άλλες ε, επιστημονικές έρευνες είτε στη βιομηχανία που είναι εξίσου σημαντικές αλλά δεν έχουν το τόσο σημαντικό λόμπι πίσω τους όπως η ε, σαρωτές μαγνητικού συντονισμού. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να έχουμε και περαιτέρω εξαιρέσεις όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, αν είναι απαραίτητο. Ε, είναι θετικό που είπατε ότι η ισότητα δεν είναι εκ της ανθρώπινης φύσης. Ο κύριος Τόμας και μετά η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε από τις επιστημονικές έρευνες έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση. Μπορώ να, να διαβεβαιώσω την κυρία Αλήν ότι και εγώ σύμφωνο μαζί της. Και εγώ. Μια φορά έπαθε ένα ατύχημα στο τένις και χρειάστηκε να μπω σε ένα μαγνητικό τομογράφο Γιατί μπαίνει, το είναι κάπως καταστροφικό, γιατί νιώθει κανείς κλειστοφοβία, πρέπει να μείνει ακίνητος και όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να κάνει κανείς κάτι αντίθετο. Όταν είναι κανείς μέσα σε αυτό το μαραφέτι όμως και ακούει την, ε, ε, τον θόρυβό του, είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό. Μπορούμε να τα αντέξουμε όλα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει αρνητικά όλους κάνει ό,τι μπορεί κανείς να είναι δυνατός να αντέξει και όλα αυτά τα πράγματα για να αντέξει την τομογραφία. Αλλά έχω καταθέσει μια άλλη τροπολογία. Λέτε ότι θέλετε να υπάρξει μια εξαίρεση για την ε, ε μαγνητική τομογραφία γιατί πρέπει και το προσωπικό να προστατεύεται. Αυτό όμως δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα το να μειώσουμε τα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών μαγνητικών τομογραφιών και αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα στους ε, ασθενείς. Υπάρχει και ο κίνητος μιας άνησης μεταχείρισης για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον τομέα αυτό. Έχω μιλήσει με πολλούς βουλευτές που είπαν και εμπειρογνώμους που είπαν ότι χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Έχουμε φυσικά πάντα εξαιρέσεις για ορισμένε περιπτώσει, αλλά μπορεί αυτό να μα οδηγήσει να έχουμε εργαζομένου πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ή μήπω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσει και τα ιατρικά κέντρα θα έχουν εξοπλισμό που να μειώνει την πραγματική ακτινοβολία για το ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει διαφορετική άποψη σε πολλά κράτη-μέλη. Στη Γερμανία υπήρξε μια συμβαστική λύση από ό,τι γνωρίζω. Εγώ έχω συζητήσει με τους συναδέλφους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες, ίσως η θέση μου να είναι μια θέση μειοψηφία, αλλά ίσως <clears throat> θα μπορέσουμε να εξετάσουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση στο τέλος. Θα χαρώ πάρα πολύ, όχι μόνο με την Ελίζαμπεθ, αλλά και με όλους τους άλλους να συζητήσω τις απόψεις. Ευχαριστώ. Ζητούμε τώρα από την Κομισιόν, από τον αρμόδιο <clears throat> διευθυντή, ο κύριος Σίλβα και ο συνάδελφός του, ποιος από τους δύο σας θέλει να λάβει το λόγο, γιατί βέβαια δεν μπορώ να έχω το λόγο να σας δώσω και στους δύο αμφί. Κύριε Σίλβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω να πω ότι θέτησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οδηγία 2012-0003. Είναι μια οδηγία που παρατείνει κατά δύο χρόνια την ε, προθεσμία για την ενσωμάτωση οδηγίας 2004-40 όσον αφορά την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έλαβε αυτή την απόφαση ούτω ώστε να αποφύγει μια γενικευμένη κατάσταση νομικής αβεβαιότητας, η οποία θα δημιουργεί το αν όταν φτάναμε στις 30 Απριλίου φέτος δεν θα είχαμε ακόμα εγκρίνει μια οδηγία για την αναθεώρηση της οδηγίας του 2004. Και υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δοθήσεις της ποικιλία των θέσεων που εκφράστηκαν σε συζητήσεις στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Πολωνικής ε, Προεδρίας. Συνεπών, δύο χρόνια θεωρούμε ότι είναι μία περίοδος εύλογη, δίνει ένα περιθώριο ασφαλείας, ούτω ώστε με σταθμισμένο τρόπο, ισορροπημένο, να ενημερωθεί και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον ενήμεροι να φτάσουμε όλοι μαζί και οι τρεις, τα τρία θεσμικά όργανα σε ισορροπημένη θέση. Σήμερα διαβιβάσαμε στο Συμβούλιο και ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σε όλες τις γλώσσες αυτή την οδηγία. Όσον αφορά την ουσία, παραμένουμε στη θέση μας, δηλαδή του Ιουνίου του 2011, που κάναμε την πρόταση αναθεώρησης. Χρειαζόμαστε ισορροπημένη οδηγία που να μπορεί να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, δηλαδή να μπορεί να παρέχει αποτελεσματική προστασία στους εργαζομένους οι οποίοι εκτίθενται στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω ενός συστήματος ας πούμε ε, εφαρμογής υποχρεωτικής οριακών τιμών στην έκθεση και ορίων προσανατολισμού και δράσεων που βοηθούν τους εργοδότες να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και διατάξεις όσον αφορά την κατάρτιση, τον ιατρικό έλεγχο και εποπτεία, τα, τις συνέπειες που έχουν τα εκνομενικά πεδία και τα μέτρα που χρειάζονται και μέτρηση αυτών. Χρειαζόμαστε όμως και μια εφαρμόσιμη οδηγία και με την εμπειρία έχουμε μάθει από το 2004 ότι κάποιες πτυχές δεν ελήφθησαν υπόψη από τους νομοθέτες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εν μέρη φέρει την ευθύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι βυθιζόμενοι σε μια οδηγία, σε μια συζήτηση που δεν λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των τελευταίων ετών, ε, ίσως χωρίς να χρειάζεται μπορούμε να καθυστερούμε την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων που είναι σημαντικά για την προστασία όλων των εργαζομένων που εκτίθενται στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στον ιατρικό τομέα, και εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις, για τους οποίους επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικέ εξαιρέσει, ελεγχόμενες προφανώς, δεν είναι μια εξαίρεση από όλη την οδηγία, αλλά εξαίρεση μόνο για την εφαρμογή των ριακών τιμών και τιμών προσανατολισμού, όμως υπάρχουν, υπάρχει σειρά μέτρων προληπτικών που προβλέπουμε για αυτούς. Πέραν αυτού υπάρχουν εκατομμύρια εργαζόμενοι που περιμένουν να προστατευτούν καλύτερα σε διάφορα κράτη-μέλη. Άρα είναι καθήκον μας να επιταχύνουμε τις εργασίες μας και τις αποφάσεις που θα λάβουμε όσον αφορά την οδηγία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σιγήτρη έχει το λόγο. Σημείωσα δεόντως όλα όσα είπαν οι σκιώδεις εισηγητές και τις ε, κατευθύνσεις και τις θέσεις που ήθελα να προβάλλουν. Λυπούμε πολύ για την αναχώρηση της Λις Λίν, που ήταν θερμή υπέρμαχος ε, της προσπάθειας και βοηθός μου ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα. Και ξέρω ότι ο στόχος που, οι στόχοι που καθορίζουμε δεν θα μπορούσαν να επιτευθούν χωρίς τη δουλειά που έκανε. Ελπίζω ότι εκεί που θα βρίσκεται να μπορέσει να συνεχίσει να μας βοηθά. Θα ήθελα να πω επίσης, όπως είπε ε, όπως υπόθηκε ότι χρειάζονται οι εξαιρέσει για τους μαγνητικούς τομογράφους. Ξέρουμε τι γίνεται στις εξετάσεις, ο καθένας έχει κάνει τις εξετάσεις. Πρέπει να επιμείνω κυρία Πρόεδρο ότι σήμερα η τεχνολογία, η χειρουργική εξελίσσεται και υπάρχουν και χειρουργικές παρεμβάσεις υψής του επίπεδου που μπορούν να γίνουν υπό έλεγχο μαγνητικών τομογράφων και σαρωτών Άρα ε, ε, βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό στάδιο εν εξελίξη. Πολύ σημαντικές εξελίξεις για τους ασθενείς είμαστε όλοι μας ε, κάποια δεδομένη στιγμή στη ζωή μας. λαμβάνω υπόψη αυτά που είπε η κυρία Ράπτη, αλλά αυτά που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη που υπάρχει να αναβληθεί, να πάει, να πάει αργότερα η, η προθεσμία ε, εφαρμογή οδηγία του 2004 διότι η προθεσμία της 21 η Απριλίου είναι σχεδόν μεθαύριο, είναι κοντά. Περιμέναμε πολύ σε αυτή την ε, Επίτροπη. Περιμέναμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταφθάσει, ούτω ώστε να μπορούμε να το συζητήσουμε. Και πολύ γρήγορα ξεκινήσαμε τη δουλειά. Ξέραμε ότι η προθεσμία ήταν πάρα πολύ κοντά. Θα συζητήσουμε μαζί στην Επιτροπή αυτή, την κοινοβουλευτική, την αναβολή της, ε, της προθεσμίας, της ημερομηνίας, Να μετατεθεί η προθεσμία, η ημερομηνία της 21ης Απριλίου, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάθε συμφέρον να μην αναβάλουμε παόριστον ε, δύο χρόνια. Σας το λέω αμέσως. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μακριά και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όλοι εδώ έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες και δείξαμε μεγάλη θέληση τόσο ώστε αυτό το κείμενο να προχωρήσει. Δύο χρόνια ήδη θα είμαστε κοντά σε μια προεκλογική εκστρατεία και ανανέωση του Κοινοβουλίου. Και πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου λογικό. Υπέχουμε ευθύνε, πρέπει να τι ανυπομιστούμε. Η κυρία Λίν μα το υπενθύμησε, διότι εργάστηκε από το 2004 πάνω σε αυτό το κείμενο. Αν θέλουμε να δώσουμε σάρκα και οστά στη δουλειά που κάνουμε, θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα από αυτό και εγώ θα προτείνω στους συναδέλφους βουλευτές όχι πάνω από ένα χρόνο για να ε, καταλήξουμε κάπου σε αυτό το κείμενο. Διότι η μη εφαρμογή της οδηγίας του 2004 είναι μη εφαρμόσιμη. Ε, το θεωρώ ότι είναι σκανδαλώδες αυτό. Με ενοχλεί τα μάλα και δεν θα ήθελα να είναι ένα κακό παράδειγμα που θα δώσουμε στους πολίτες μας, δηλαδή να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι ικανή να οργανωθεί με θετικό τρόπο και για να προστατεύσει τους εργαζομένους της, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσει και τους ασθενείς. Θα κάνω ό,τι μπορώ και θα κινητοποιηθώ δεόντως για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, σκιώδεις συγκητές, για τη δουλειά που έκανα πάνω σε αυτό το θέμα και περιμένω ακόμα περισσότερα στις διαπραγματεύσεις που θα έρθουν, ούτω ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ κυρία Συγκήτρια. Λοιπόν. Θα προσθέσουμε λοιπόν στο ημερολόγιό μας, σύμφωνα με αυτά που θα πούν και οι συντονιστές και συντονίστριες, και έτσι θα ψηφίσουμε βασικά στις 13 Φεβρουαρίου σε έκτακτη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο. Τώρα, όσοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής, ούτε υπάλληλοι της ομάδας, να φύγουν από την αίθουσα να την εγκαταλείψουν γιατί τώρα θα συνεδριάσουμε και κλεισμένων των θυρών. Μπορείτε να πιείτε ένα κοκτέιλ απ' έξω, αλλά Παρακαλώ ηρέμωσα.